Καθίστε παρακαλώ, θα χρειαστείτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω ισπανικά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε όλοι και όλες. Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σήμερα Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού θα βρίσκεται μαζί μας μία ομάδα νέων, επικεφαλής νέων του Σουδάν, βρίσκονται στην τελευταία σειρά της αίθουσας και θα παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας σήμερα το πρωί. Τους καλωσορίζω και τις καλωσορίζω θερμά, τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Έχουμε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα όπως πάντα σήμερα το πρωί και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με την εξέταση των θεμάτων που αποτελούν προτεραιότητα για τη δουλειά μας. Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του τράφικιν στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να επιμείνει κανείς το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων, το τράφικιν, είναι η δουλεία του 21ου αιώνα λέγεται. Εγώ λέω ότι είναι δουλεία γενικότερα γιατί ίσχυε και τον 21ο αιώνα και τον 20ο και τον 19ο, τον 18ο και τον 17ο. Είναι δουλεία, τελεία και παύλα, και το μόνο που γίνεται είναι να εξυγχρονίζουν τις μεθόδους τους οι, αυτοί οι οποίοι κάνουν τράφικινγκ. Ουσιαστικά για δουλεία πρόκειται γιατί μιλούμε για αγορά και για πώληση ανθρώπινων όντων προκειμένου να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Εμπλήρη απουσία της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Για να προσεγγίσουμε λοιπόν αυτό το περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει χίλιες οπτικές γωνίες και χίλιες διαφορετικές διαστάσεις, θελήσαμε να έχουμε ένα πάνελ υψηλής ποιότητας, της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και θα σας παρουσιάσουμε τους παρεμβαίνοντες κάθε φορά που θα παίρνουν το λόγο ο καθένας. Καταρχάς, έχουμε τον κύριο Σεμπαστιάν Βολ, ο οποίος είναι ερευνητής και αναλυτής στο γραφείο, το Περιφερειακό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την δράση συνεργασίας ε, κατά της εμπορίας ανθρώπων, κατά του τράφικιν. Είναι το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών που έχει την έδρα του στη Μπανκόγκ, UN Act λέγεται, και θα μας μιλήσει για τις διαφορετικές κατηγορίες αυτού του φαινομένου. Καλημέρα σας κύριε Μπολ, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, σας ακούμε. Good morning and thank you, Madam Chair. Um, I trust that Καλημέρα σας ε, κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε. Είναι τιμή για εμάς ε, την ε, UNACT, την συνεργασία του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και για μένα προσωπικά που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή την ακρόαση. συνεδρίαση αυτή αφορά την εμπορία ανθρώπων που ουσιαστικά πρόκειται για την ε, πρόσληψη, μεταφορά, η διατήρηση ανθρώπων σε μορφές ε, βαριάς εκμετάλλευσης ε, μέσω μέσων απατηλών και μου έχετε δώσει ε, μου έχετε αναθέσει κάτι το σχεδόν αδύνατο σε 10 λεπτά να σας παρουσιάσω το παγκόσμιο μέγεθος του προβλήματος. Δεν είναι μόνο αδύνατον λόγο του χρόνου, αλλά επειδή η αλήθεια είναι πως η λαθρέα φύση του εγκλήματος ε, αλλά και οι διαφορές στους ορισμούς ε, και άλλοι παράγοντες ε, το καθιστούν ε, πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσουμε την εμπορία ανθρώπων, ειδικά στο παγκόσμιο επίπεδο. Γίνονται όμως κάποιες ε, προσπάθειες και νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως μία από τις πιο συστηματικές προσπάθειες είναι η εκτίμηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την καταναγκαστική εργασία και η Μπεάτα Ανδρέας νομίζω είναι εκεί πέρα σήμερα μαζί σας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις σχετικές ε, δημοσίευσεις. Η ακριβής ε, σχέση βεβαίως ε, μεταξύ των δύο είναι κάτι το συζητήσιμο, αλλά συνδέονται στενά σε μεγάλο βαθμό και αλληλεπικαλύπτονται. Οπότε οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ουσιαστικά θεωρούνται χοντρικά ότι δίνουν μία εικόνα για την εμπορία ανθρώπων. Αυτό το οποίο βγήκε το 2012 είναι πως μιλάμε για 20,9 εκατομμύρια ανθρώπους σε καταναγκαστική εργασία ανα πάσα στιγμή κατά μέσο όρο τα 10 χρόνια που μας πέρασαν. Πάνω από τα 14 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους ήταν σε συνθήκες εκμετάλλευσης της ε, καταναγκαστικής εργασίας, 68% του συνολίνου. 4,5 εκατομμύρια ήταν σε συνθήκες σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Και εδώ πέρα αυτό είναι κάτι το σημαντικό που θα ήθελα να το πω. Νομίζω πως ε, δικαιολογείται μια ευρύτερη παρέμβαση πέρα από την ε, συνήθη συζήτηση που συχνά αφορά μόνο τη σεξουαλική εκμετάλλευση και να ασχοληθούμε και με την εκμετάλλευση της εργασίας. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κατά τις εκτιμήσεις ε, του ILO ε, είναι πάνω από το 50% των περιπτώσεων αυτών και η ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μεκόγκ εδώ πέρα που δρούμε εμείς δηλαδή, ξεκινώντας από την Κίνα στο βορρά, ε, Βιετνάμ, Λάος, Μιανμάρ, Καμπότζη και Ταϊλάνδη, έχει τις πιο εκτεταμένες ροές ε, καταναγκαστικής εργασίας και εμπορίας ανθρώπων. Και θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή γιατί αντιλαμβάνομαι πως ε, θα υπάρξει και μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εστιαστεί στην Νοτιοανατολική Ασία. Όταν μιλάμε λοιπόν για την περιοχή του Μεκόγκ, ε, είναι πολλές περιπτώσεις. Καταναγκαστική εργασία στον τομέα της αλληλείας, ε, βιομηχανία, κατασκευές, ε, οικιακή εργασία, αναγκαστική γάμη, ακόμα και αφαίρεση οργάνων. δεδομένου του περιορισμένου χρόνου θα ήθελα να τονίσω δύο τάσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Η μία, η οποία νομίζω είναι ενδιαφέρουσα επειδή είναι καινούρια και η άλλη που είναι ενδιαφέρουσα γιατί αφορά άμεσα την Ευρώπη. Η πρώτη είναι η καταναγκαστική γάμη ε, προς την Κίνα και εντός της Κίνας. Αυτό σχετίζεται με την πολιτική του ενός παιδιού και την προτίμηση των Κινέζων για τα αγόρια που έχει οδηγήσει σε πλεόνασμα ανδρών, το οποίο το 2020 θα είναι 45 εκατομμύρια. Αυτό έχει καταλήξει σε μια ζήτηση για συζύγους και σεξουαλικές υπηρεσίες, γυναίκες συζύγους που και πάλι έχει καταλήξει στην ε, καταναγκαστική ή απατηλή στρατολόγηση γυναικών εντός της Κίνας αλλά και ε, πιο μακριά ε, για να τις πάνε στην Κίνα με σκοπό και το γάμο μεταξύ των άλλων. Βλέπουμε σε γειτονικέ χώρες, ειδικά στο Μιανμάρ και στο Βιετνάμ, κάποιες τέτοιε τάσει. αλλά βλέπουμε τέτοια πράγματα και από πιο μακριά, όπως είπα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, από χώρε όπως η Καμπότζη. Το πλεόνασμα αυτό είναι κάτι το ανησυχητικό λόγο των επιπτώσεων και οι κινέζικες αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν ε, το πρόβλημα και να συνεννοηθούν και με τους λοιπούς ε, εταίρους. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω σήμερα το πρωί αφορά την περίπτωση της, ε, του αλευτικού κλάδου της Ταϊλάνδης. Η Ταϊλάνδη είναι μεγάλος εξαγωγές ελευθερικών προϊόντων και εξάγει και στην Ευρώπη. Ο κλάδος απασχολεί 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και ε, πάρα πολλούς ε, μετανάστες. Ε. Πολλοί από αυτούς είναι μη καταγεγραμμένοι. Συχνά από χώρες όπως η Μιανμάρα, το Λάος και η Καμπότζη. η εξάντληση των ηχθειοποθεμάτων στον κόλπο της ε, Ταϊλάνδης ε, σημαίνει πως τα σκάφη βγαίνουν όλο και πιο έξω στη θάλασσα και μένουν ε, στα ανοιχτά ακόμα και χρόνια μερικές φορές. Επίσης, πρόκειται για σκληρή εργασία βεβαίως η Αλία και σε συνδυασμό με τους μακρόχρονους πλώες αλλά και τον αυξημένο ανταγωνισμό στην βιομηχανία έχει κάνει την εργασία σε αυτόν τον κλάδο ε, πάρα πολύ δύσκολη και αποθητική για τους Ταϊλανδούς αλλά και για τους μετανάστες που ενημερώνονται από τις κοινότητες τους για τις συνθήκες που επικρατούν. Ως αποτέλεσμα αυτού καταφεύγουν ε, συχνά οι εργοδότες ε, σε μέσα απατηλά ή καταναγκαστικά. Είχαμε πρόσφατα και ένα ρεπορτάζ του Associated Press που τόνισε τις συνθήκες ξυλοδαρμία, ακόμα και φόνος έγινε. Βεβαίως ε, η εφοδιαστική αλυσίδα είναι πολύ πλοκή και είναι δύσκολο να ξέρουμε από πού έρχονται τα προϊόντα και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να φτάνουν σε ευρωπαϊκές αγορές προϊόντα καταναγκαστικής εργασίας. Η κυβέρνηση της Θαϊλάνδης επίσης έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και το θεωρεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Και έχει κάνει κάποια πρώτα βήματα. Κατέγραψε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες εργαζόμενους. Ζήτησε και από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία και από τη δική μας την υπηρεσία ε, και άλλες υπηρεσίες που βοηθούν την κυβέρνηση της Ελλάδας. Αλλά ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα και στο να έρθουμε σε επαφή με Ευρωπαίους, γι' αυτό σήμερα σας μιλάω, μεταξύ των οποίων και αντιπροσωπείες ε, στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και με μονομένες κυβερνήσεις ε, και με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί νομίζω πως και ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη έχει ένα ρόλο να παίξει. Νομίζω λοιπόν ότι τα 10 λεπτά που μου δώσατε πέρασαν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και αναμένω περαιτέρω συζήτηση την ώρα που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. 10 λεπτά ακριβώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μείνετε ή πρέπει να φύγετε. Ευχαρίστω να μείνω. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπεάτε άντρε ειδική διευθύντρια για το ειδικό πρόγραμμα δράσης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας η οποία θα μας μιλήσει για το ποιος κερδίζει από αυτό το φαινόμενο, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος από το UNACT ε, με πολύ ωραίο τρόπο σας παρουσίασε τα δεδομένα σχετικά με το εύρος ε, του, των δραστηριοτήτων ε, trafficking. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις λύσεις και πρέπει να πω ότι μου αρέσει αυτός ο καταμερισμός εργασίας. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο μέρος της παρουσίασής μου θα ήθελα να σας δώσω ακόμα μερικές πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις βασικές οικονομικές αιτίε και τα όσα ξέρουμε για την οικονομική πλευρά του, της καταναγκαστικής εργασίας και στο δεύτερο μέρος να εστιάσω, όπως είπα, στις λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να σας πω πώς έχουν τα στοιχεία παγκοσμίω. Όπως είπε ο συνάδελφος, η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν 21 εκατομμύρια άντρε γυναίκες και παιδιά σε καταναγκαστική εργασία που είναι αντικείμενο ε, τράφικινγκ για καταναγκαστική εργασία και ε, και της ε, ε, σεξουαλικής Αυτή είναι μια εκτίμηση ε, βέβαια. Ε, ε, δεν έχουμε εθνικά στοιχεία ε, για να έχουμε μια πιο αξιόπιστη παγκόσμια εκτίμηση και πρόσφατα ξεκινήσαμε μια μελέτη για να έχουμε πιο αξιόπιστη στοιχεία όσον αφορά την συχνότητα του φαινομένου. Ας έρθουμε όμως στην οικονομική πλευρά της καταναγκαστικής εργασίας. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το εμπόριο ανθρώπων είναι ε, μια πολύ ε, μεγάλη δραστηριότητα η οποία ε, δημιουργεί 150 δισεκατομμύρια σε παράνομα κέρδη το χρόνο. Τα δύο τρίτα των κερδών αυτών δημιουργούνται στην βιομηχανία του σεξ. Όμως η πλειονότητα των 20 αυτών εκατομμυρίων ανθρώπων είναι αντικείμενο εκμετάλλευση σε χαμηλά αμοιβόμενου τομεί τη οικονομίας όπως είναι ε, η γεωργία, η αλία, οι οικοδομές, η βιομηχανία και η οικιακή εργασία. Ε, η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 880.000 γυναίκες, άντρες και παιδιά που είναι αντικείμενο εμπορίας με τον σκοπό ε, την καταναγκαστική εργασία ή δουλεύουν σε συνθήκες σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όλο αυτό βέβαια ε, το, φαινόμενο υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ε, διάφορων οικονομικών ε, κλάδων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν είναι μόνο big business αυτό, είναι πολύ κακό για τους εργαζόμενους και δημιουργεί τεράστιο κόστος για τις κοινωνίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της καταναγκαστικής εργασίας και του τράφικινγκ. Έλλειψη εσόδων σε σε, σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παραδείγματος χάρη. Το εμπόριο ανθρώπων βλέπουμε ότι όλο και πιο πολύ ε, σχετίζεται με ε, παγκόσμιες αλυσίδες προσφοράς. Αναφέρθηκε το παράδειγμα του ελευτικού στόλου της Ταϊλάνδης που ε, τραβάει την προσοχή τώρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια είδαμε το φαινόμενο και σε άλλους οικονομικούς τομείς όπως τη ε, ε στην ε, βιομηχανία ενδυμάτων ε, και ηλεκτρονικών. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη σε όλη την αλυσίδα προσφοράς. Ο κίνδυνος είναι λοιπόν να παραπλανηθούμε ως προσθετίες και να αυξηθεί το φαινόμενο της αναγκαστικής εργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ελληνική διακυβέρνηση της ε, ε, αγοράς εργασίας ε, των μεταναστών που πολλοί από αυτούς είναι υπερχρεωμένοι σε μια αλυσίδα ιδιωτών διαμέσων. Όταν έχουν χρεωθεί για να μεταναστεύσουν οι μετανάστες αυτοί είναι πολύ πιο πιθανό να καταλήξουν σε καταναγκαστική εργασία. Η παράνομη και άτυπη στρατολόγηση δημιουργεί δισεκατομμύρια κερδών ε, και στις χώρες προέλευσης και στις χώρες προορισμού. Η ε, παγκόσμια ολοκλήρωση των ε, οικονομιών μας δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για πολλούς και έχει συμβάλει σε αύξηση του πλούτου σε πολλές περιοχές του κόσμου, αλλά επίσης δημιουργεί ευκαιρίες για αυτούς που αναζητούν το, εύκολο και παράνομο κέρδος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς διαφεύγουν. Ε, δεν πληρώνουν για τα εγκλήματά τους, διότι είναι ε, ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστεί η νομοθεσία σε ε, διασυνοριακό διακρατικό επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα αυτού, μόνο λίγα θύματα ε, μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τα όσα έχουν ε, υποφέρει. Τι πρέπει να γίνει. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την νομοθεσία. Πέρυσι οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων ε, στο ILO ε, υιοθέτησαν ένα δεσμευτικό ε, πρωτόκολλο το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση του 1930 για την καταστική εργασία του ILO και την σχετική σύσταση. Ο σκοπός είναι ιδιαίτερα να ενισχυθεί η πρόληψη, η προστασία και τα ένδικα μέσα, διορθωτικά μέσα. συμπληρώνοντας το σχετικό πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι αυτά τα νέα μέσα που διαθέτουμε για να εμποδίσουμε την αλυσίδα αυτή της καταναγκαστικής εργασίας. Το πρώτο ε, ε, σημείο είναι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ε, το πρωτόκολλο και η συζήτηση τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι αιτίε, ε, η ρίζα του κακού. Αυτό απαιτεί επενδύσεις στην κοινωνική προστασία και στην εκπαίδευση, ιδίω σε βάλλοντα νοικοκυριά που συχνά είναι αποκλεισμένα από τα υπάρχοντα συστήματα προστασίας. Ε, πολύ συχνά η πρώτη γενιά των μέτρων κατά του τράφικινγκ εστίαζε στην ε, ε, ποινικοποίηση, στην εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων και την δίωξη. Αυτά τα μέσα ήταν φυσικά πολύτιμα, αλλά είναι καιρός πλέον να αναπτύξουμε αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης που σχετίζονται με την διακυβέρνηση της αγοράς εργασίας και την ε, μετανάστευση. Δεύτερον, πρέπει να ε, εξισορροπηθούν οι επεμβάσεις που αφορούν αφενός την προσφορά και αφετέρου τη δίδυση. Και πάλι η πρώτη γενιά των μέτρων κατά του τράφικινγκ μερικές φορές δυσανάλογα δεν την έμφαση στην ε, προσφορά παρά στην ζήτηση όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Είναι όμως πάρα... Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθούν δυνατότητες τα ε, ε, θύματα του τράφικινγκ, εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί ε, έμφαση στην πλευρά της ε, ζήτησης ε, για φτηνή εργασία και υπηρεσίες. Και πάλι το παράδειγμα του ελευθερικού στόλου της Ταϊλάνδης είναι ένα καλό παράδειγμα. Το πρωτόκολλο και η σύσταση του ILO καλούν και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να ενισχύσουν την παθήπνησή τους ε, για να ε, μετριαστεί ο κίνδυνος καταναγκαστικής εργασίας. Ε, οι διατυπώσεις αυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα επιχειρηματικά και ανθρώπινα δικαιώματα. πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και πέραν αυτού. Ε, κάποια κράτη ε, πρόσφατα ε, υιοθέτησαν νομοθεσία που επιβάλλει στις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν ε, τις πληροφορίες για το εμπόριο ανθρώπων. Ε, τα μέτρα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν από ισχυρή νομοθεσία όσον αφορά την επέκταση των εξουσιών των επιθεωρητών εργασίας ιδιαίτερως. Και τέλος, ε, ας μιλάμε για εργαζόμενους και όχι για θύματα. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται σε καταναγκαστική εργασία δεν έχουν απαχθεί από κακούς ε, αφεντάδες. Παρόλο που δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια τραγικά ε, φαινόμενα στις σημερινές κοινωνίες. Όμως τα περισσότερα θύματα του τράφικινγκ αρχικά συνένεσαν στη στρατολόγηση για την απασχόλησή τους. Είναι εργαζόμενοι και ε, αναζητούν μια αξιοπρεπή εργασία πολύ συχνά είναι μετανάστες εργαζόμενοι μακριά από το σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενδυναμωθούν. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα και όχι να διασωθούν. Το πρωτόκολλο και η σύσταση του ILO ε, περιλαμβάνουν μέτρα που θα αποσκοπούν ε, το όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στα ένδικα μέσα, ανεξάρτητα από, ε, από το νομικό καθεστώς τους, ε, βάσει του οποίου βρίσκονται ε, σε μια χώρα. Πρέπει να τονιστεί, αυτό τονίζεται σε όλες τις ε, διατάξεις του ILO, ε, η, τονίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένδικα μέσα. υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μπορέσουν να οργανωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι θύματα του τράφικινγκ και της καταναγκαστικής εργασίας. δεν υπάρχει τίποτα πιο ε, ισχυρό από την συλλογική ε, δράση των ανθρώπων αυτών. Ε, υπάρχει λοιπόν μια νέα στρατηγική ε, του ILO για την αποτελεσματική ε, εξάλληψη του τράφικινγκ. Ε, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστούν γρήγορα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρκέτα Όγκροβα, Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Οργάνωσης που καταπολεμά το τράφικινγκ. Θα μας μιλήσει για την υπεράσπιση και τα δικαιώματα των θυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Είναι τιμή για μένα που μιλώ εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση σε ανθρώπους που εκπροσωπούν τόσο σημαντικά θεσμικά όργανα ε, στην καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων. Η Λαστράντα είναι ε, μια οργάνωση ομπρέλα που στεγάζει 8 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και εγώ εργάζομαι στο γραφείο της Τσεχίας. Πριν από αυτό εργαζόμουν σε άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτή η προοπτική με ενδιαφέρει η προοπτική των σημάτων ως ανθρωπίνων όντων, ως άτομα των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται και καταστρατηγούνται. Έχω μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μου, θα πρέπει λοιπόν να παραμερίσω όλα όσα έχω γράψει στην παρουσίασή μου και να τονίσω μόνο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει πολύ ε, μεγάλα βήματα σε επίπεδο νομοθετικών βημάτων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των γυναικών, υπήρξε μια ανάπτυξη ε, ε, θεσμικών διατάξεων. Έχουμε έγγραφα όπως το πρωτόκολλο κατά του τράφικιν των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το θέμα αυτό, έχουμε σχετικές οδηγίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα αυτά τα έγγραφα τα δικαιώματα των θυμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο. Είναι η προσέγγιση με το θύμα στο επίκεντρο. Ε, δεν μας εκπλήσει αυτό το οποίο θα έρθει Δυστυχώς δεν δουλεύουμε μέσα σε ένα χρυσό πύργο, αν θέλετε, σε έναν ιδεατό κόσμο. Πολύ συχνά η προσέγγιση του θύματος στο επικεντρό αντιβαίνει ή αντιφάσκει με άλλα νομοθετικά κείμενα και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Π.χ. οι πάροχοι υπηρεσιών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν διαφωνία έναντι των δικαιωμάτων των εκμεταλλευόμενων ανθρώπων. Η προσέγγιση με το θύμα στο επίκεντρο που σημαίνει ότι όλα γυρίζουν γύρω από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων είναι σε αντιπαράθεση με την προσέγγιση της ποινική δικαιοσύνης. Μπορούν αυτές οι δύο προσεγγίσεις να συμβαδίσουν, ωστόσο σε άλλες στιγμές της ζωής ε, του θύματος τράφικιν η εισαγγελική προσέγγιση της ποινική δικαιοσύνης ουσιαστικά ε, υπερβαίνει τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων του τράφικιν γίνονται σεβαστά ανεξαρτήτως του αν συνεργάζονται με την εισαγγελία την ποινική δικαιοσύνη ή όχι. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα αυτά και είναι πολύ θεμητός και λογικός ο φόβος των θυμάτων αυτό που νιώθουν εάν ή όταν δεν συνεργάζονται με την αστυνομία. και σε κάποιο βαθμό μπορεί τα θύματα αυτά να τα χρησιμοποιεί ή να τα εκμεταλλεύεται ε, και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση αυτή η, η εισαγγελία, η ποινική δικαιοσύνη προκειμένου να πετύχει το στόχο της και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Δεν θα πρέπει το θύμα να βρίσκεται σε μια κατάσταση κατά την οποία απειλείται η ζωή του ή είναι σε ευπαθή και πιο ευαίσθητη και πιο ε, προβληματική κατάσταση από αυτή στην οποία βρισκόταν πριν ε, αναφερθεί και πριν ε, καταθέσει στην αστυνομία. Τελευταία έχουμε όλο και πιο κατασταλτική προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης με συγκεκριμένη στόχευση υπηκόων συγκεκριμένων τρίτων χωρών. Βλέπετε λοιπόν ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των θυμάτων τράφικιν από τις πολύ αυστηρές ε, και κατασταλτικές ε, μεταναστευτικές πολιτικές. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μία των θυμάτων και από την άλλη των πολιτικών εθνικής ασφάλειας σε περιπτώσεις ε, οποιασδήποτε απειλής τοπικής, εθνικής ή διεθνούς ευρωπαϊκής υιοθετούνται οι πιο επίγουσες διατάξεις για την ασφάλεια και έτσι καταστέλλεται η όποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περικόπτονται τελικά όλα αυτά τα δικαιώματα με αόρατο τρόπο θα έλεγα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αντιφάσεις, αυτές οι δύο-τρεις αντιφάσεις τις οποίες σας παρουσίασα ε, μεταξύ της προσέγγισης που έχει το θύμα στο επίκεντρο και ε, τα υπόλοιπα θεμητά ε, συμφέροντα των κρατών μελών. Νομίζω ότι για να λύσουμε αυτές τις αντιφάσεις πρέπει να υιοθετήσουμε μια συνολική, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της νομοθεσίας και κατά διάρκεια της σύλληψης και διατύπωσης της νομοθεσίας αυτής θα πρέπει η νομοθεσία και το νομοπαρασκευαστικό έργο σε οποιοδήποτε πεδίο να μην ε, παρεμποδίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά ή θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο ε, της εξέτασης οποιοδήποτε κειμένου στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Παραδείγματα που δείχνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας και μετά της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Πρώτον, ταυτοποίηση των θυμάτων τράφικιν, των ατόμων. Οι διατάξεις είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Η ενσωμάτωση αυτών των διατάξεων έχει γίνει πολύ σωστά και υπάρχουν εθνικοί μηχανισμοί που αντικατοπτρίζουν αυτές τις διατάξεις και όσοι ε, εργάζονται σε αυτό το τομέα ειδικοί εμπειρογνώμονες είναι πολύ καλά καταρτισμένοι και πολύ καλά εξειδικευμένοι. Το βασικό πρόβλημα είναι η έγκαιρη ταυτοποίηση στο, στη γραμμή πυρός, στη γραμμή του μετόπου αν θέλετε, δηλαδή από πλευράς αστυνομικού, του πρώτου που βλέπει αυτό το θύμα. Το όργανο της τάξης που βλέπει πρώτο αυτό το θύμα ε, στερείται γνώσεων για να μπορέσει να ταυτοποιήσει ε, ότι πρόκειται για ένα θύμα trafficking και έτσι μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής. Στη, στη δουλειά μας ένα παράδειγμα. Μία πελάτησα ήρθε από την Ιταλία, ήταν θύμα trafficking, είχε μεταφερθεί από την Αφρική στην Ιταλία και είχε πλαστό διαβατήριο. Την πιάσαν στα τσεχικά σύνορα και... και και και την κατηγόρησαν ότι πήγε παράνομα στην Απικράτεια. Και κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα τη συμβαίνει και τώρα που αποθήθηκε στην Ιταλία και θα είναι πάλι θύμα τράφικη. Έχουμε επίσης μια περίπτωση τριών εργαζομένων, διάσημη στην Ευρώπη περίπτωση, στη Τσεχία πάνω, των 150, ε, πάνω από 150 εργαζόμενοι ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης στον τομέα της υλοτομίας. Η Λαστράντα ε, τους βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους και παρακολουθούμε πέντε χρόνια την εξέλιξη των ποινικών και προανακριτικών διαδικασιών. Τελικά, ποτέ δεν εξετάστηκε το θέμα αυτό υπό τη σκοπιά του τράφικιν. Και πάντοτε το αίτημα αυτό απορρίπτεται για λόγους διαδικαστικούς, για λόγους τυπικούς και ούτου καθεξής. Μετά από πέντε χρόνια το Τσεχικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφαίνεται τώρα για την ε, παραβίαση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη ε, βάσει και της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης για την υποχρέωση να διώκονται όλες οι περιπτώσεις τράφικιν από πλευράς θητών και θα υπάρξει και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τίθενται λοιπόν ερωτήματα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Είναι λόγω έλλειψη γνώσεων, είναι λόγω αδυναμίας ταυτοποίηση των θυμάτων, υπησέρχονται άλλοι παράγοντες που θέλουν να στρέψουν το παιχνίδι προ όφελό του. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση. Έρχομαι τώρα στο θέμα τη αποζημίωση. Είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα ε, των θυμάτων, αλλά είναι και το πιο δύσκολο να το ασκήσει κανείς. Πρώτον, λόγω έλλειψης ε, πληροφόρησης από πλευράς ε, των ατόμων που υφίστανται τράφικιν, τέτοιου είδους διατάξεις είναι γνωστές στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αυτές δεν έχουν πολύ μεγάλη δυναμικότητα, δεν μπορούν να έχουν πολύ πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα άτομα, άρα η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών δεν είναι επαρκείς, οι δικηγόροι και η λειτουργοί των δικαστικών αθουσών γενικότερα δεν γνωρίζουν γι' αυτό το δικαίωμα για αποζημίωση και πολύ συχνά το δικαίωμα αυτό περιορίζεται λόγω άλλων ε, καταστάσεων, όπως είναι για παράδειγμα η ε, αδυναμία του ατόμου να παραμείνει στη χώρα μέχρι ότου αποφασιστεί το θέμα της αποζημίωσης ή επειδή δεν ε, είναι νομίμως διαμένων το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μία από τις εγγυήσεις αυτό, ότι δηλαδή θα προστατεύουμε τα δικαιώματα των ατόμων που υφίστανται τράφικιν σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ε, των λοιπόν στοιχείων. Ίσως η διατύπωση είναι πολύ ήπια. Λέει ότι τα κράτη-μέλη shall be entitled Δηλαδή δεν είναι δεσμευτικά. Λέει ότι τα κράτη-μέλη θα δικαιούνται να μην ασκούν διώξει για διάφορε παραβάσει έναντι των ατόμων τα οποία είναι θύματα τράφικιν. Αυτή είναι μια πολύ ήπια διατύπωση. Και δεν υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να μην ασκήσουν διώξει προκειμένου να μην καταστρατηγηθούν τα ατομικά δικαιώματα των ατόμων που εμπλέκονται σε τράφικιν, των θυμάτων. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση με το θύμα στο επίκεντρο είναι πολύ σημαντική και μπορώ να σας δείξω παραδείγματα που δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοστεί, υπάρχει σε κείμενα και μάλιστα ε, το αποτέλεσμα είναι πολύ επιτυχημένο. Μιλούμε για θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων τράφικιν και είναι προϋπόθεση ε, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων τράφικιν. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα συνεργαστούν με τον εκάστοτε εισαγγελέα οι αστυνομικέ αρχές ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ούγκροβα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζωή Σακελιάδου πολιτική βοηθό της κυρίας Βασιλιάδου η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Συντονίστρια για το θέμα αυτό η οποία την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να είναι ε, μαζί μας. Θα ακούσουμε όμως εσάς. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Εκπροσωπώ σήμερα την ε, κυρία Βασιλιάδου, συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της εμπορίας ανθρώπων που για κάποιους λόγους, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε ε, να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και για το ότι διατηρείτε το ζήτημα ανοιχτό. Λίγα λόγια για την έντολη και τον ρόλο της ε, συντονίστριας. Πρόκειται για ένα άρθρο στην σχετική οδηγία, το νομικό μέσο το οποίο ορίζει το νομικό πλαίσιο εντός της Ένωσης και άρα έχει εντολή να συντονίζει και να δίνει στρατηγικές κατευθύνσεις εντός ε, της Ένωσης, ε, των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αλλά και εξωτερικά. Και μάλιστα από τον τίτλο ήδη της ακρόασης αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος εδώ πέρα είναι η εξωτερική διάσταση της εμπορίας ανθρώπων και το πώς το λαμβάνουν υπόψη οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καλύτερο νομίζω θα ήταν να σας έκανα μια παρουσίαση στην αρχή της ευρωπαϊκής διάστασης και προσέγγισης σε σχέση με την εξωτερική δράση. Τέλος πάντων, θα το κάνω τώρα. Η εμπορία ανθρώπων ε, είναι μαρίτατη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σοβαρό έγκλημα, διεθνές έγκλημα που δεν μπορεί καμία χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της. Η εμπορία ανθρώπων είναι, όπως σωστά είπε η Πρόεδρος, αφορά την πώληση και αγορά ανθρώπων και υπηρεσιών. Μιλάμε για ανθρώπους. Και βεβαίως το θέμα είναι και τα κέρδη και η ζήτηση. Συχνά ακούμε για ευάλωτους ε, ανθρώπους ε, κάτι το οποίο συνεισφέρει αλλά δεν προκαλεί την εμπορία. Υπάρχει ζήτηση και κέρδος που δημιουργεί το φαινόμενο και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Τώρα, η εμπορία ανθρώπων απαγορεύεται ρητά από την χάρτα θεμελιδών δικαιωμάτων. Στο άρθρο 5 και πρέπει να τονίσουμε πως ε, η απαγόρευση αυτή προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και εφαρμόζει το πρωτογενές δικαίου της Ένωσης. Επίσης, σχετικές ε, διατάξεις υπάρχουν στις συνθήκες ε, της Ένωσης ε, στα κομμάτια που αφορούν την κανονική μετανάστευση και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύντο χρόνο κατάφερε να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικό και θεσμικό το οποίο εστιάζεται στα θύματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει μια διεπιστημονική προσέγγιση ένα πλαίσιο το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ λεπτομερές στο τι συμβαίνει εντός της Ένωσης αλλά και στην εξωτερική διάσταση Λοιπόν, δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζουμε την πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιολογεί τις προσπάθειες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με την σχετική οδηγία και θα δημοσιεύσουμε και την πρώτη έκθεση συμμόρφωσης της ε, σχετικής ε, οδηγίας και πώς εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη σημειώστε πως Απρίλιο του 2013 ήταν η προθεσμία μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο και αυτή τη στιγμή δύο κράτη-μέλη μόνο μας έχουν ενημερώσει για μερική μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο. Όπως έχετε ίσως ακούσει, η Κομισιόν έχει δύο σημαντικά θέματα, την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Ατζέντα και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα της Ασφάλειας και βέβαια η Συμπορία ανθρώπων είναι σημαντικό μέρος Πράγματι το θέμα αφορά και τη μετανάστευση και έχει μια παγκόσμια διάσταση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το εσωτερικό και την εσωτερική, την εξωτερική διάσταση. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Δεν θα χρησιμοποιήσω εκτιμήσεις αλλά στατιστικά δεδομένα για την περίοδο 2010-2012 καταγράψαν 30.146 θύματα εμπορίας ανθρώπων ε, τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Βεβαίως αυτό δεν είναι η πραγματική κατάσταση και έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. Τα θύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί 65% των καταγεγραμμένων θυμάτων είναι πολίτες της Ένωσης, αλλά οι πολίτες τρίτων χωρών προέρχονται από την Ιγυρία, τη Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Βιετνάμ και Ρωσία. Κάποιοι από αυτούς ε, τους ανθρώπους ε, μπήκαν ε, με τρόπο παράνομο ή με κάποιον άλλο τρόπο και χρειάζεται εδώ πέρα να είμαστε σαφείς για τις έννοιες και τους όρους όπως εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τη σύνδεση, αλλά μιλάμε για διαφορετικά ζητήματα. Συχνά τα συγχαίουμε και πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε σαφείς ως προς αυτό. Τώρα, η πρόληψη βεβαίως ε, έχει μεγάλη σημασία και θα ήθελα εδώ πέρα να επαναλάβω πως η νομοθεσία της Ένωσης ε, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν την εμπορία ανθρώπων και την ζήτηση που οδηγεί σε αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης με διάφορα μέσα. Η εξωτερική διάσταση ε, βεβαίως ε, είναι κλειδί. Όπως ε, ξέρετε είχαμε το σχετικό έγγραφο του 2009 το οποίο είχε αντικατασταθεί από τη στρατηγική της Ένωσης ε, για την εμπορία ανθρώπων η οποία ξεκαθαρίζει πως η εμπορία αυτή είναι βασικό κομμάτι σε όλους τους διαλόγους με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επανέλθω με λεπτομέρειες. Το Δεκέμβριο του 2012 το Συμβούλιο θέτησε μια λίστα χωρών προτεραιότητας με τις οποίες επιθυμεί να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες προτεραιότητας περιλαμβάνουν την Αλβανία, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Μαρόκο, την Ιγυρία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Ουκρανία και το Βιετνάμ. Οι περιφέρειες περιλαμβάνουν τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, τις ε, χώρες της ε, Καρικόμ, ε, το δρόμο του μεταξιού, την Κεντρική Αφρική κτλ η χρηματοδότηση παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια. Πολλά έργα έχουμε χρηματοδοτήσει, όλα αυτά τα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει την πολιτική και θα δει όλη την υπάρχουσα χρηματοδότηση γιατί πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και να δούμε το τι γίνεται, τι δεν γίνεται και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Η επανεξέταση πολιτικής είναι κάτι το παραδοτέο όπως λέμε. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ανοίξει διαγωνισμός ε, και μέχρι σήμερα περιμένουμε υποβολές προτάσεων. Ο ρόλος ε, τώρα της εμπορίας ανθρώπων αναφέρεται σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως παγκόσμια προσέγγιση στη μετανάστευση και την κινητικότητα της ε, συνεργασίες κινητικότητας Μαρόκο, την Ισία και τα λοιπά που επίσης λαμβάνουν υπόψη ε, την εμπορία. Επίσης είναι στοιχείο στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κάνουμε με πολλές ε, χώρες όταν μιλάμε για περιφερειακό διάλογο με την Αφρική και τη διαδικασία του Ραμπάτ και εκεί πέρα αναφέρεται το ζήτημα αυτό μπορεί να έχετε ακούσει τη λεγόμενη διαδικασία του Χαρτούμ και εκεί πέρα προτεραιότητα η εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με την Υπουργική Δήλωση. Η κοινή ατζέντα για τη μετανάστευση με την Ιγυρία επίσης αναφέρει την εμπορία ανθρώπων και η διαπραγμάτευση με τη Βραζιλία επίσης θα καταλήξει μια συμφωνία που θα περιέχει τέτοια στοιχεία. Η Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθερότητας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Επίσης ε, το περιέχουν αυτό το στοιχείο. Η πολιτική γειτονία, η ανατολική εταιρική σχέση, όλα αυτά. Σημαντικότερο, έχουμε την κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως είναι ίσως εταίρος κοινωνία των πολιτών. Ακόμα και η νομοθεσία της Ένωσης αναφέρεται στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε χρηματοδοτήσει μια σειρά έργων. Το πιο πρόσφατο ήταν ένα τριετές έργο σχεδόν 11 εκατομμυρίων ευρώ στην ε, Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελίνου για να οικοδομηθεί δυνατότητα σε τρίτες χώρες, ε, δικαιώματα μεταναστών, οργανώσεις που τα προωθούν και συμπεριλαμβανομένων και των ε, οικιακών βοηθών. Όλα αυτά είναι στην σελίδα μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ένα πολύ καλό πλαίσιο, αλλά τώρα πρέπει να δούμε το τι γίνεται. Το εάν εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο και να αξιολογήσουμε τα... ποια ήταν τα επιτεύγματά μας. Και να πω πως ε, εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους, για αγορά και πώληση ανθρώπων και υπηρεσιών. Έτσι η ευθύνη είναι ακόμη πιο επιτακτική πλέον. Τώρα, αν θέλετε να μου κάνετε και ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους που θα μοιραστούν μαζί μας τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τις ερωτήσεις. Και μετά θα δώσουμε πάλι το λόγο στους ομιλητές ε, του πάνελ. Αν υπάρχει χρόνος. Η κυρία Οστροβίτσιος, παρακαλώ. Ο κύριος Οστροβίτσιος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτό το, αυτή τη συνεδρίαση. Εκτιμώ ιδιαίτερως τις πληροφορίες που λάβαμε από τις διαφορετικές πηγές, από τα μέλη του πάνελ. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ στη συλλογή των στοιχείων και στην ταυτοποίηση, την αναγνώριση των θυμάτων, την καταχώρηση και παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, δεν ε, χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένα νούμερα. Ουσιαστικά χανόμαστε στη διαδικασία. Η στρατηγική που υιοθετήσατε το 2000, η στρατηγική που η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2011 αναφέρει ότι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλογή δεδομένων είναι σημαντική και τα αποτελέσματα αναμένονται το 2014. Έχετε περισσότερε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Υπάρχουν επιτεύγματα και αν ναι, ποια είναι αυτά και τι μένει να γίνει ακόμα. Και δεύτερον, κάποιος από το πάνελ θα μπορούσε ίσως πιο συγκεκριμένα να απαντήσει στο εξής. Με διαφέρει η διοικητική δυναμικότητα των αρχών επιβολής του νόμου, που υποτίθεται ότι είναι επιφορτισμένες με το καθήκον να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό. Σε ποιο βαθμό βλέπετε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, καλύτερη γνώση, παραδοχή, δυνατότητα αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου από πλευράς κρατών μελών. Σε ποιο βαθμό βλέπετε να υπάρχει, αν υπάρχει αυξημένη διασυνοριακή, ε, διεθνική συνεργασία έτσι ώστε να υψωθεί πραγματικά ένα φράγμα ε, που ε, θα αποτρέψει αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είχα ορισμένες ερωτήσεις να κάνω στους καλεσμένους μας. Ξέρουμε ότι ένα από τα πιο διαδομένα και επικερδή διεθνή φαινόμενα είναι το εμπόριο ανθρώπων. Είναι βιομηχανία που εκτιμάται σε 150 δισεκατομμύρια δολάρια και αφορά διάφορα άτομα είτε στο ε, αφορά την ε, εργασία ανηλίκων, παραδείγματος χάρη, σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η κρίση όσον αφορά την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για την καταπολέμηση του φαινομένου. Ε, αν ε, χρειάζονται νέε παρεμβάσει σε σχέση με τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί ε, αναφέρομαι παραδείγματο χάρη και σε φορολογικούς ελέγχους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η αντίθεση ε, από την ποινική σκοπιά ανάμεσα στο θύμα και στον θήτη. Γιατί τα θύματα πολύ συχνά ε, υφίστανται ε, ποινικέ διώξεις και ποινές. Ε, αναφέρομαι ιδίως σε γυναίκες μετανάστριες σε ορισμένες χώρες υπάρχουν πραγματικά παράδοξα φαινόμενα ως προς αυτό. Αυτό συνδέεται και με την ε, τρίτη μου ερώτηση που αφορά την ε, αρρωγή και την προστασία των θυμάτων. Δεν υπάρχει αυτό πάντα. Αντίθετα, ε, σπάνια έχουν την απαραίτητη βοήθεια ε, τα θύματα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, τα παιδιά ιδίω και οι ανήλικοι. Ε, κατά τη γνώμη σας είναι απαραίτητο να γίνει βάθηση προ την κατεύθυνση αυτή. Και τέλος, μία πληροφορία. Ε, θα ήθελα. Η κυρία Άντερς μίλησε για αυτό το θέμα. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει ένα κάποιο είδος συνδικαλισμού. Ε, δεν ξέρω αν ε, ε, ε, ήρθατε σε επαφή με τα παραδοσιακά συνδικάτα, τη CGI, παραδείγματος χάρη. Και αν η επαφή αυτή σας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι κεντρικός ο ρόλος του συνδικαλισμού. Και αν έχετε συνεργασία μαζί τους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το θέμα ε, παλιό αλλά και πρόσφατο είναι ε, ένα θέμα για το οποίο τα συνδικάτα έχουν πολλά να προσφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λαχμπίλερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν εδώ και μας παρουσίασαν πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι ακρόαση για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά κυρίως δίνει το ενδιαφέρον της την εσωτερική διάσταση του θέματος ενώ η δική μας υποεπιτροπή είναι μέρος της εξωτερικής οικογένειας. Με αυτά ασχολούμαστε. Τώρα, ως προς την εκπρόσωπο της συντονίστριας, μιλήσατε για τις χώρες προτεραιότητες σας. Βλέπετε καμία προσαρμογή δική τους Ίσως θα πρέπει να προσταθούν και άλλες χώρες, αυτές τις χώρες προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ε, να γίνουν βελτιώσεις. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και δεύτερον, ο κύριος Παντσέρη αναφέρθηκε στην ανάγκη του να δώσουμε προσοχή στην ευαλωτότητα των παιδιών που είναι θυμάτων τράφικιν. Θεωρείται εμπόριο αυτό το πράγμα, εμπορία το πρώτο μισό του 2015 θα υπάρξει αξιολόγηση αυτής της ε, δραστηριότητας. Μέχρι που έχετε φτάσει, μπορείτε να μας πείτε. Και εσείς, κυρία Μπεάτε Άντερς, στη, στη δική σας παρουσίαση είπατε ότι πρέπει να κάνουμε τα θύματα να αποκτήσουν ισχύ, να πάρουν την, ε, τη δύναμή τους στα χέρια τους και γι' αυτό δεν θα πρέπει τόσο να μιλούμε, να, ε, να λέμε ότι είναι τόσο θύματα όσο το ότι είναι εργαζόμενοι και θέλουν να βελτιώσουν ε, την κατάστασή τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Όμως τα παιδιά πώς εντάσσονται σε αυτή τη συλλογιστική σας. Από εκεί και πέρα η έκθεση στην οποία αναφερθήκαν οι παριστάμενοι δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές της Ασίας, μιλάει και για τη Βραζιλία. Θέλουμε μια παγκόσμια άποψη. Ε, αναφέρομαι στον κύριο Σεπάστιαν Μπολ ε, που μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Όμως τα περισσότερα θύματα του τράφικιν είναι στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πώς μπορούμε αυτά να τα ε, ταιριάξουμε μαζί. Και ο κύριος Αυστρεπίτσιος το, το ρώτησε αυτό τι κάνουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ε, πώς έχουν ε, καταφέρει να συνδυάσουν αυτό με την καταπολέμηση του τράφικιν. Υπάρχουν επιτυχίες. Εσείς κυρία Μπρόκοβα λέτε ότι δουλεύετε ε, στην μπροστινή γραμμή, τη γραμμή του πυρός μαζί με τη Frontex. Πώς εφαρμόζουν λοιπόν το, την καταπολέμηση του τράφικιν εκεί στα σύνορα, επί τόπου, εκεί που υπάρχουν τα προβλήματα, έχουν την απαραίτητη οργάνωση, την απαραίτητη ε, εκπαίδευση. Και σίγουρα εκτός εκακροάσεις θα σας θέσουμε πολύ περισσότερες ερωτήσεις. Ωστόσο, να δω λίγο τις σημειώσεις μου αν έχω ξεχάσει κάτι, γιατί μάλλον ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, βέβαια, είχα ερωτήσεις που τις έχουν ήδη κάνει οι συνάδελφοι, δεν τις επαναλαμβάνω. Ναι, Έχετε εμπειρία για το πόσο πολύ οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες προτεραιότητας, πόσο συμμετέχουν, πόσο ασχολούνται. Αν δείτε ας πούμε για τις χώρες που εντάσσονται στη συνεργασία, ε, τις χώρες του κόλπου, συνεργασία με τις χώρες του κόλπου, ε, Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει διαφορετικά ή να αναλάβει περισσότερες δεσμεύσεις. Πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Λοχμπίλερ, λέει η Πρόεδρος. Σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να ε, συζητήσετε με την κυρία Λοχμπίλερ, η οποία είναι η συγγήτρια της σχετικής έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Σίγουρα η κυρία Λοχμπίλερ θα συνεχίσει, θα χρειάζεται να συνεχίσει τη συνεργασία με εσάς, τους εμπειρογνώμονες, τις εμπειρογνώμονες και ειδικού που είναι μέλη του πάνελ. Επομένως θα έχετε την ευκαιρία όλη την εβδομάδα να ανταλλάξετε απόψεις. Ο κύριος Δεμεσμέκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις. Πολλές ε, ερωτήσεις έχουν ήδη γίνει και έχω κάποια επιπλέον σχόλια για κάποιες ερωτήσεις και εγώ και αν δεν έχετε αντιρρήσει θα συνεχίσω στη γλώσσα μου που είναι τα Ολλανδικά. Ε, ε, το εμπόριο ανθρώπων όπως και η κλιματική αλλαγή και η τρομοκρατία είναι ένα διασυνοριακό φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον καρκίνο της εμπορίας ανθρώπων με μεγάλο συντονισμό της επιτήρησης των συνόρων, ε, της αστυνομίας, ε, των δικαστηρίων. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα νομοθετικά μέσα που υπάρχουν, τα μέσα που έχουμε, τις γραμμές χρηματοδότησης, ε, βεβαίως ε, τα ζητήματα ετέθησαν. Ε, πρέπει να αξιολογήσουμε τι γίνεται, πρέπει να δούμε ποια μέσα έχουμε και ποια από αυτά λειτουργήσαν καλύτερα. Ποια μέσα είναι τα πιο αποτελεσματικά. Αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε. Ένα τρίτο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και κινητικότητα στα σύνορά μας τα νότια αλλά και τα ανατολικά προβλήματα, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπετε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την ροή και Μήπως μπορούμε να κινηθούμε πιο προληπτικά Και τελευταίο ερώτημα, πώς πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για ενημέρωση του δικού μας ε, πληθυσμού. Τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε, νομίζω ποιον ρόλο βλέπετε για εμάς σε αυτή τη ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στις ε, προσκεκλημένες μας για να απαντήσουν. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω το ε, κύριο Σεμπαστιάν Μπόλ, ο οποίος και αυτός είναι εμπειρογνώμων και μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Να σας ρωτήσω, κύριε Σεμπαστιάν Μπόλ, για τα δύο πιο καινούργια ζητήματα Πρώτον, τους ε, καταναγκαστικούς και υποχρεωτικούς γάμους, στην Κίνα κυρίως, και δεύτερον, διακίνηση, εκμετάλλευση, εμπορία εργαζομένων στην, ε, στον κλάδο των αλλιευτικών βιομηχανιών επεξεργασίας αλλιευμάτων, ε, που τελικά τα προϊόντα τους παίρνουν ευρωπαϊκή σφραγίδα. Έχετε περισσότερα στοιχεία Ξέρω ότι δεν μπορείτε να μας τα πείτε όλα, δεν έχουμε και χρόνο άλλωστε, όμως με ενδιαφέρει ιδιαίτερος ο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την παρουσία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες ωφελούνται από αυτή την κατάσταση μεταναστών εργαζομένων που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευση στον, στην αλληλευτική βιομηχανία, ε, στην Κίνα και με ενδιαφέρει και το θέμα των υποχρεωτικών καταναγκαστικών γάμων στην Κίνα. Δεν ξέρω αν ακολουθούν τα ίδια κυκλώματα με τα κυκλώματα που ακολουθεί η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση ή αν είναι νέα κυκλώματα που δημιουργούνται. Εν πάση περιπτώσει αυτά τα δύο θέματα με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Εμένα ως πρόεδρος τη υποεπιτροπή αυτή, γιατί δεν, τα, δεν γνώριζα πολύ καλά πώ έχει αυτή η κατάσταση. Ε, κύριε Μπόλ, είστε ακόμα μαζί μας, μπορείτε να παραμείνετε, μπορείτε να μας απαντήσετε. Εάν συμφωνείτε και μπορείτε να ε, παραμείνετε, ξεκινούμε ε, με την τελευταία ομιλήτρια η οποία θα απαντήσει πρώτη. Ευχαριστώ. Good question. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις καλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες και θα ξεκινήσω από την τελευταία παρατήρηση που είπε η συγγήτρια κατάλογος χωρών και περιοχών προτεραιότητες. Αυτό ήταν μέρος των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που όντως ανέφεραν ότι σε τακτικά διαστήματα θα πρέπει να επανεξετάζεται η λίστα αυτή. Τώρα, ε, τούτου λεχθέντος θα πρέπει όντως να επανεξετάσουμε και τις προτεραιότητές μας από αυτή την άποψη. Ε, όπως είπα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λύγει το 2016. Είναι λοιπόν καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει και ποια θα είναι η στρατηγική μας μετά το 2016. Η δουλειά που κάνουμε στην εξωτερική διάσταση του εμπορίου ανθρώπων είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζουμε στενά τη δράση μας με την ε, ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με άλλες υπηρεσίες και επίσης κινητοποιούμε και τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες είτε έχουν υψηλή προτεραιότητα είτε όχι. Και από αυτή την άποψη η δουλειά της αντιπροσωπείας μας επί τόπου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ευαλωτότητα των παιδιών είναι ένα μεγάλο ζήτημα που επίσης έχει εντοπιστεί ως τέτοιο από την Europol. Με χαρά μου μπορώ να σας πω ότι ε, εργαζόμαστε δραστήρια προς την κατεύθυνση αυτή. Έχω φέρει εδώ κάποια αντίτυπα το βρίσκονται στην είσοδο. Το 2004 η Επιτροπή, Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημιούργησε έναν οδηγό για τα παιδιά που δεν ε, τυχάνουν χάνουν ε, φροντίδας. Το εγχειρίδιο αυτό έχει μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει πληροφορίες και εμπειρίες από λειτουργούς ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Και το προωθούμε συνεχώς. Ένα άλλο θέμα είναι το δικαίωμα, τα δικαιώματα των θυμάτων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα άτομα αυτά ψάχνουν μια καλύτερη ε, ζωή αλλά είναι θύματα ενός φρικτού εγκλήματος και υπό την ιδιότητα αυτή έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε διάφορα προστατευτικά μέτρα που υπάρχουν για αυτούς. Ε, έχουμε ε, ανάγκη από ε, μια συνολική παρουσίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων σε μια γλώσσα και με, τρόπο έκφρασης που να είναι προσβάσιμος για ε, τα θύματα, αλλά και ε, που θα προωθηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Μας ρωτήσατε για τη μελέτη που πραγματοποιούμε ε, σχετικά με τα παιδιά ως ομάδα υψηλού κινδύνου. Ε, σύντομα η μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί, θα είναι διαθέσιμη και θα έρθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τι κάνει για το θέμα αυτό. Μόλις δούμε τι αποδίδει και τι όχι, ως ε, ε, θεματοφύλακες της ηθικής θα κάνουμε την πρώτη ε, έκθεση συμμόρφωσης το 2015, όπου θα αξιολογούμε πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόσουν την ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία σε εθνικό επίπεδο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θύχθηκε ε, αφορά τις ε, δυνάμεις επιβολής του νόμου. Και τι γίνεται εκεί. Πολλά γίνονται και πολλά αποδίδουν. Η Europol είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό ε, εφαρμόζει τα δικά της προγράμματα, ε, το impact όπως λέγεται, το τράφικινγκ ε, αποτελεί προτεραιότητα και παραμένει προτεραιότητα για την Europol και σε τακτά διαστήματα ενημερωνόμαστε για τις σχετικές διαδικασίες. Πιστεύουμε όντως ότι θα ήταν επικοδομητικό να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση των κρατών μελών για να προωθήσουμε τη δουλειά που κάνουν μπορώ να σας πω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις από καθημέλη έχουν υποφεληθεί από τα προγράμματα αυτά και από τη χρηματοδότηση που διατίθεται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ταμείο των Συνόρων. Είναι διαθέσιμα. Ε, έχουμε δύο στοχευμένα ε, σεμινάρια για το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής. Ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα που δείχθηκε είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ε, ένας πολύ βασικός παράγοντας. Η Κομισιόν το έχει μάθει αυτό με πολύ σκληρό τρόπο. Δημοσιεύσαμε δύο έγγραφα εργασίας, η Eurostat δηλαδή, δημοσίευσε δύο έγγραφα εργασίας για το ε, εμπόριο ανθρώπων. διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η συλλογή συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Ε, θα πρέπει να ε, είναι ε, πιο τεκμηριωμένες οι πολιτικές μας. Αλλά ακόμα και για ένα σήμα, ένα να υπάρχει, έχουμε ηθική και νομική υποχρεώση να δράσουμε. Ε, συμβάλλουμε λοιπόν, συμβάλλουμε στις διαδικασίες ε, συλλογής δεδομένων και έχουμε χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα που προωθούν την ευρωπαϊκή διάσταση στη συλλογή δεδομένων. Όλες αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην ε, μεσοπρόθεσμη έκθεση για τη στρατηγική και ε, υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές και στη σχετική ιστοσελίδα. Τέλος, μία παρατήρηση σχετικά με το ρόλο των ε, εργασιακών ενδιάμεσων και το, τις σχετικές παρατηρήσεις. Σε συνεργασία με τον οργανισμό του Δουβλίνου μελετάμε τον ακριβή ρόλο των ενδιάμεσων για εργασιακά θέματα όσον αφορά το τράφικινγκ. Η μελέτη αυτή θα είναι επίσης διαθέσιμη κατά τους προσεχείς μήνες. Και επίσης ε, θα ξεκινήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Συνεργασία κατά του τράφικινγκ ε, όπου η καλή πλευρά της επιχειρηματικότητας ε, θα προσπαθήσει να προωθήσει μια μορφή επιχειρήσεων που δεν θα βασίζεται στο τράφικινγκ και στην καταναγκαστική εργασία. Δεν μιλάμε για εταιρική ευθύνη μιλάμε για νομική ε, ευθύνη των επιχειρήσεων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο ε, στο εμπόριο ανθρώπων. Και τέλος, οι οικονομικές έρευνες είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια όπως ακούσαμε ε, κερδών από το τράφικινγκ. Πρέπει τα χρήματα αυτά να τα ανοιχνεύσουμε, να τα παρακολουθήσουμε. Η Europol ε, κάνει τις σχετικές έρευνες και σύντομα θα μάθουμε περισσότερα από αυτού. Πάντως είναι ένας ε, τομέας ε, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Marketa uh, thank you for the... Ευχαριστώ, Μαρκέτα Χρόνκοβα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Δεν θα αναφερθώ σε όλες, γιατί κάποιες απαντήθηκαν και υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές λοιπόν. Το ένα αφορά το ζήτημα της ε, ποινική έρευνας, ε, της αυτοποίησης και το θέμα βέβαια των διοκτικών αρχών πρέπει να πούμε πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος κάθε χρόνο, τουλάχιστον στις χώρες που παρακολουθούμε υπάρχουν περισσότερες καταδίκες ή έρευνες για την εμπορία ανθρώπων. Και δεν νομίζω πως ε, είναι επειδή αυξάνεται ο όγκος, απλά γιατί γίνεται καλύτερη η ε, ταυτοποίηση. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο κενό γιατί πολύ απλά ε, βεβαίως ε, είναι πολύ, πάρα πολλά τα άτομα ε, που είναι αντικείμενο εμπορίας σε σχέση με τις έρευνες και τις καταδίκησεις. Κάτι άλλο, για να καταδικαστεί κάποιος, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο για τα δικαστήρια και τους εισαγγελείς. Οπότε, τι βλέπουμε συχνά, επιμερίζεται το έγκλημα σε μικρότερα δικήματα Δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον ε, η βεβαιότητα ότι θα καταδικαστεί κάποιο για απάτη, σωματική βία κτλ. Γιατί όλες αυτές οι πτυχές τη εμπορία ανθρώπων μπορεί να μην ε, υπάρχουν ε, και δεν είναι σίγουρη η καταδίκη. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό το οποίο πρέπει να δούμε. Βεβαίως υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπα, της ταυτοποίησης όχι μόνο στα σύνορα της Ένωσης, ε, όλοι όσοι είναι στην πρώτη γραμμή που έρχονται σε επαφή ε, με άτομα που δυνητικά είναι αντικείμενο εμπορίας δεν ειδοποιούνται εγκαίρως, ε, συχνά επαναπατρίζονται είτε στη χώρα από όπου ξεκίνησαν είτε στη χώρα προέλευσης και θα πρέπει να υπάρχουν αυτό το οποίο η οδηγία λέει κάποιες ομάδες που θα ταυτοποιούν αυτούς τους ανθρώπους και θα γίνει βέβαια και με τους ανθρώπους ε, που πέφτουν ε, στη θάλασσα. Τώρα το θέμα των συνδικάτων ε, δυστυχώς νομίζω πως είναι γνωστό σε πάρα πολλές χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ. Τα συνδικάτα έχουν πρόβλημα φήμης θα έλεγα, δεν πιστεύει κανείς ότι εργάζονται για το καλό των εργαζομένων. Είχαμε κάνει ένα πανευρωπαϊκό πάνελ και προσκαλέσαμε και τα τσέχικα συνδικάτα και μία από τις δηλώσεις που έγινε ήταν πως ε, εμείς ε, δεν θέμε τους μετανάστες να γραφτούν στα συνδικάτα, ε, εμείς τα θέμε για τσέχους. Βλέπετε λοιπόν πως υπάρχει τεράστια διαφορά ε, όσον αφορά την ανάπτυξη των συνδικάτων σε διάφορες ε, χώρες ε, και στην δικιά μας την περιφέρεια θα χρειαστούν μία ή δύο γενιές για να δούμε οργάνωση των εργαζομένων όπως βλέπουμε στη Λατινική Αμερική ή αλλού. Και τέλος η πρόληψη. Η πρόληψη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο όμως στην πλευρά των ε, ανθρώπων, αλλά οπωσδήποτε στην πλευρά των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, τη λεγόμενη πλευρά της ζήτησης. Όσο η ζήτηση καθορίζεται μόνο από τη φτηνή εργασία, δεν θα προχωρήσουμε καθόλου στην πρόληψη. Και όσον αφορά στην πρόληψη στην πλευρά των ε, πιθανών ανθρώπων που είναι αντικείμενα εμπορίας ε, ακόμα και αν γνωρίζουν τους κινδύνους ζουν πολλοί από αυτούς σε τέτοιες συνθήκες που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο και να πάνε αλλού ακόμα και αν το ξέρουν το τι θα γίνει οπότε πρέπει να δούμε και τις ρίζες ε, τις αιτίες του προβλήματος δηλαδή τέλος για τη μεταχείριση των θυμάτων σε σχέση με τη μεταχείριση των παραβατών. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα αγρόκτημα μαριχουάνας όπου συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις εκμεταλλεύονται ε, ανθρώπους ε, σε άθλιες ε, συνθήκες, τους έχουν περιορισμένους και είχαμε μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ήταν έγκλειστος επί μήνες του περνούσαν φαΐ από ένα παράθυρο και παρόλα αυτά κατέληξε στο ίδιο κελί με τους ανθρώπους που τον είχαν κρατούμενο και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Δηλαδή, άμα τον έχουν εκεί πέρα έγκλειστο, νομίζω είναι προφανές ότι δεν πήγε εκεί εθελοντικά. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε τα θύματα, οι μετανάστες, από τους δράστες. Και να είναι σαφές πώς πρέπει να μην τιμωρούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεάτε Άντρες. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με κάποια ζητήματα που αφορούν τους ορισμούς, γιατί το είπε και η κυρία Λοχμπίλερ, αλλά και τα θέματα των δεδομένων σχετίζονται με το πώς χρησιμοποιούμε τους νομικούς ορισμούς. Κατ' ουσίαν έχουμε τρία πράγματα στο διεθνές δίκαιο. Εμπορία ανθρώπων, ε, καταναγκαστική εργασία το τραφικίνγκ. Ε, είναι διακριτά όλα αυτά, αλλά υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη. Η πρόεδρος είπε πως πρόκειται για σκλαβιά. Η εμπορία ανθρώπων και σκλαβιά είναι το ίδιο. Ε, υπάρχουν αποχρώσεις στον νόμο. Κοιτάξτε, η καταναγκαστική εργασία είναι κάτι το ευρύτατο. Κατ' ουσίαν ε, αφορά το στοιχείο του καταναγκασμού. Αλλά τα στατιστικά αν αλλάξουμε τους ορισμούς θα είναι και υψηλότερα. Θα είναι υψηλότεροι αριθμοί. Πρέπει δηλαδή να βάλουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους ε, στην περίπτωση της ε, καταναγκαστικής εργασίας υπηρεσιών. Και θα έχουμε μετά και διαφορετικές προτεραιότητες. Δηλαδή, αν δούμε τα νούμερα, τα περισσότερα θύματα είναι σε καταστάσεις ε, παραδοσιακής ε, καταναγκαστικής εργασίας. Ε, κάποιοι μετανάστευσαν, αλλά όχι απαραίτητα. Κάποιοι γεννήθηκαν σε αυτή την κατάσταση και μετά βεβαίως το θέμα αφορά και τα παιδιά. Υπολογίζουμε πως 5,5 εκατομμύρια του συνόλου είναι παιδιά ανήλικοι. Και τα παιδιά οι νέοι, όπω λέμε, χειρότερε συνθήκε εργασία πρέπει να διασωθούν και να προστατευτούν. Αλλά δεν σημαίνει πώ θα πάνε στο σχολείο μετά. Γιατί κάποια από αυτά είναι σε νόμιμη ηλικία για να εργαστούν. Οπότε θα πρέπει να εργαστούν ακόμα και αν σταματήσει η καταναγκαστική εργασία. Και αυτό έλεγα ουσιαστικά τα περισσότερα θύματα αναζητούν εργασία. Γι' αυτό ε, έκαναν συχνά επικίνδυνα ταξίδια και βεβαίως ε, χρειάζονται και εισόδημα ακόμα και όταν βγουν από αυτή την κατάσταση. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις διάσωσης που βλέπουμε. Βεβαίως τα παιδιά πρέπει να τα δούμε διαφορετικά και αυτό υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και έρχομαι άρα στο επόμενο θέμα, αν επαρκεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετική οδηγία της Ένωσης, όπως ξέρετε, βασίζεται στην ε, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο Διεθνές Δικαίο και άρα ε, είναι αρκετά υψηλών προδιαγραφών ε, παγκοσμίω με την υιοθέτηση νέου πρωτοκόλου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Μπορούμε να δούμε κάποιες από αυτές τις διατάξεις ξανά όπως είπα στο νέο πρωτόκολλο, έχουμε πολύ καινοτόμες ε, διατυπώσεις για το ρόλο των επιχειρήσεων και την επιμέλεια που πρέπει να δείχνουν τα ζητήματα των συνδικάτων. Το 2005 το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ξεκίνησε αυτό το οποίο λέμε την Παγκόσμια Συμμαχία κατά της καταναγκαστικής ε, εργασίας και συνεργαζόμαστε στενά με συνδικάτα στον τομέα των κλαδικό σε επίπεδο παγκόσμιο και εθνικό και η Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, έχει σχηματίσει ένα δίκτυο ε, επαφών ε, των συνδικάτων για περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε τώρα του εποπτικού Βλέπουμε τώρα ένα υποπτικό σύστημα του ILO λόγω ακριβώς ε, του ενισχυμένου ρόλου των συνδικάτων. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει κάποια έργα που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και των ΜΚΟ και υπάρχει νομίζω ένα έργο που συνεχίζεται και κάποιες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα ανταλλαγούν φέτος. Οπότε υπάρχει σαφώς ένας ρόλος που ε, μπορεί να παίξει, ο οποίος ε, πρέπει να ενισχυθεί. Νομίζω πως υπήρχε άλλο ένα ερώτημα για τις ε, διοκτικές αρχές, το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω. Συμφωνώ με άλλους όταν λένε πως υπάρχει σαφώς μια αύξηση στην κατανόηση των διοκτικών αρχών για το τι εστί εμπορία ανθρώπων και πως το διακρίνουμε από άλλες περιπτώσεις ή από κακές ε, συνθήκες εργασίας ε, ή από το λαθρεμπόριο. Αυτό το οποίο απαιτείται λοιπόν είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες ε, για αυτό το θέμα. Π.χ. επιθεώρηση εργασίας αλλά ουσιαστικά η καλύτερη εργασία, συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, ε, της επιθεώρησης εργασίας ε, και των ε, αρμοδίων για τη μετανάστευση. Έχοντας πάντα κατά νου πως η επιθεώρηση εργασίας δεν θα πρέπει βεβαίως να έχει στόχο να επιβάλλει την νομοθεσία περί μετανάστευσης γιατί μπορεί έτσι να υπάρξει πρόβλημα για να την εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι. Αυτά. Σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ και τώρα ο Σεβάστιαν Πόλ από την Βαγκόγκ. Ευχαριστώ. Ακούω τον εαυτό μου, λέει ο μιλτής. Ε, ε, χαίρομαι που έγινε αυτή η συζήτηση για την σαφήνεια των ορισμών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες και έννοιες. Θα συμφωνήσω όμως με την Πεάτε Άντρες ότι ιδιαίτερα όσον αφορά ε, το ανθρώπινο εμπόριο και την καταναστική εργασία υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση αυτών των φαινομένων, αλλά η συζήτηση ακόμα κρατάει ε, και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτή την ε, ε, θεωρητική συζήτηση και άκουσα και για την επερχόμενη έκθεση και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η σχέση ανάμεσα στο τράφικινγκ και την καταναγκαστική εργασία που θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο στην Μπαγκόγκ ε, αυτό σχετίζεται και με μια ερώτηση που μου έγινε σχετικά με τους καταναγκαστικούς γάμους. Το φαινόμενο αυτό επίσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ιδίως σε σχέση με τον ορισμό του ε, εμπορίου ανθρώπων, διότι ο γάμος καθ' αυτός δεν θεωρείται ότι είναι εκμετάλλευση. Το ερώτημα λοιπόν ε, είναι σε ποιο σημείο γίνεται εκμετάλλευση ο γάμος. Ίσως η χρήση βίας είναι κάτι που το προσωμιάζει με το τράφικινγκ. Εδώ αυτό που είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη αυτά που σα εξήγησα νωρίτερα, είναι σημαντικό, σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο καταναγκαστικό γάμο κατά κανόνα συμπεριλαμβάνει και κάποια μορφή σεξουαλική εκμετάλλευση καθώ επίση και καταναγκαστική ε, εργασία παραδείγματο χάρη είναι καταναγκαστική οικιακή εργασία στα, στα σπίτια και σεξουαλική εκμετάλλευση ε, διότι όπως είπα προηγουμένως ε, τίθεται το όλο ζήτημα της ε, γεννήσης παιδιών από τις γυναίκες αυτές που παντρεύτηκαν με αυτόν τον καταναγκαστικό τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν μορφές εκμετάλλευσης ε, σεξουαλικής και εργασιακής. Πράγμα που ε, ε, μπορεί να εντάξει το φαινόμενο του καταναγκαστικού γάμου στο ευρύτερο φαινόμενο του εμπορίου ανθρώπων, του τράφικινγκ. Ε, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση πάντως του φαινομένου διότι δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς και από τις κινητικές αρχές. Ε, έχουμε διάφορους εταίρους ε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε ε, για την διερεύνηση αυτού του φαινομένου των θυμάτων που μεταφέρονται με σκοπό τον καταναστικό γάμο από την Καμπότζη προς την Κίνα. Εξετάζουμε το φαινόμενο από διάφορες οπτικές γωνίες. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για ποιο σκοπό ε, προορίζονται ή έχουν μια ιδέα αλλά είναι διαφορετική από την ε, πραγματική προοπτική που τους περιμένει, δηλαδή τον καταναστικό γάμο. Σε άλλες περιπτώσεις ε, ξέρουν ότι τελικά πρόκειται να παντρευτούν, αλλά οι συνθήκες αποδεικνύουν ότι είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που τους έχουν υποσχεθεί. Αυτές είναι διάφορες πτυχές της εκμετάλλευσης λοιπόν και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά. Και αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω αυτό το σημείο είναι πολλές χώρες, επειδή υπάρχει ε, αυτό το φαινόμενο και αυξάνεται από ό,τι φαίνεται, έχουν ε, υιοθετήσει κάποιες πολιτικές που ε, αναχαιτήσουν τη μετανάστευση και γίνονται πολλές ε, συζητήσεις σχετικά με το ότι, για παράδειγμα, οι μόνες γυναίκες δεν θα επιτρέπεται να ταξιδέψουν προς την Κίνα εκτός αν καταθέσουν μια εγγύηση ή ε, ότι δεν θα ε, παντρευτούν αλλοδαπούς ε, Ηλικία πάνω από ένα όριο ή με περιουσία κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Ε, υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις λοιπόν από τις χώρες της περιοχής σαν απάντηση στο φαινόμενο αυτό που περιγράφουμε. Κάποια από αυτά τα μέτρα όμως κατά πάσα πιθανότητα προκαλούν περισσότερη ζημιά παρά διορθώνουν τα πράγματα. Δεδομένης δε της κλίμακος του φαινομένου των ε, ανήπαντρων, δηλαδή ανδρών που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή στην κοινωνία της Κίνας και δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού τους, ε, το πρόβλημα αυτό γίνεται πολύ σοβαρό. Τώρα, για τον αλληλευτικό τομέα. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που μπορεί να βρει κανείς εύκολα ε, μια έρευνα του Associated Press που δημοσιεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα και όπου γινόταν λόγος ιδιαίτερα για ένα νησί της Ινδονησίας ε, ε, όπου διάφορα θύματα καταναγκαστικής εργασίας ε, βρήκαν καταφύγιο ε, αφού ε, δραπέτευσαν από ε, αλληλευτικά σκάφη στα οποία δούλευαν καταναγκαστικά στα ανοιχτά της θάλασσας. Μια άλλη έρευνα είναι του Guardian και σχετίζεται περισσότερο με τη βιομηχανία γαρίδας και πώς στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού πολλά παρεπίπλατα αλλιεύματα, δηλαδή ε, ψάρια τα οποία ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση και στα πλαίσια της καταναγκαστικής εργασίας ε, οδηγούνται στην ε, διατροφική αλυσίδα σε βιομηχανίες γαρίδας. Ε, και τα προϊόντα αυτά καταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό στις ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης μια σχετική έρευνα έκανε και το BBC πέρυσι. Επιπλέον και εμείς έχουμε δημοσιεύσει ε, ε, εδώ για την αλληλευτική δραστηριότητα της περιοχής ΖΟΑΕΛΑΟ δηλαδή, δημοσίευσε πέρυσι μια έκθεση για ολόκληρο τον αλληλευτικό τομέα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Ε, η προσέγγιση μας είναι ε, συνεργατική και συλλογική και γι' αυτό ε, στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε υλικό που προέρχεται από πολλές πηγές και από όλους τους εταίρους μας και αφορά το τράφικινγκ σε όλη την περιοχή. Επίσης, όπως έλεγα προηγουμένως, η Κίνα και το Βιετνάμ ίσως θα έπρεπε να είναι χώρες προτεραιότητας στις ε, προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των ε, εξωτερικών της ε, σχέσεων. γιατί οι δύο αυτές χώρες έχουν στενές σχέσεις με διάφορους εμπλεκόμενους και ίσως θα μπορούσαν να διευκολύνουν. Ένα τελευταίο σημείο γιατί αναφέρθηκε, το θέμα των ε, διοκτικών αρχών και η Μπεάτε νομίζω το είπε αυτό, ότι η ενδυνάμωση των εργαζομένων και των μεταναστών εργαζομένων μεταξύ αυτών είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή δράση των ε, διοκτικών αρχών ε, στον εντοπισμό μορφών εκμετάλλευσης. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά στη δικιά μας περιοχή υπάρχουν περιορισμοί ε, όσον αφορά ε, την ε, συμμετοχή σε συνδικάτα και λοιπά και γενικά το να, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς ανοιχτά για συνθήκες εκμετάλλευσης που υφίσταται χωρίς να υποστεί συνέπειες. Υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, λοιπόν, αλλά και θέμα ε, προθυμίας αυτών που είναι θύματα εκμετάλλευσης να έρθουν και να συνεργαστούν με τις διεκτικές αρχές για τέτοια θέματα. Και αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας κλειδί ε, στις προσπάθειές μας να ακουστούν περισσότερες τέτοιες ιστορίες. Ε, ευχαριστώ όλους εσάς. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις αντιδράσεις και τα σχόλια. Η κυρία Πρόεδρος βγήκε από την αίθουσα, γι' αυτό και προεδρεύω εγώ εδώ και λίγα λεπτά. Έχουμε κακά νέα. Μαθαίνουμε ότι στην Τσεχία πρέπει να περιμένουμε να έρθει η επόμενη ή και μεθεπόμενη γενιά για να μπουν στα συνδικάτα ε, οι μετανάστες. Μαθαίνουμε ότι τα ευρωπαϊκά ψάρια είναι ύποπτα και πρέπει να υφίστανται ελέγχους. Όλο δεινά είναι τα νέα που έρχονται. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ όλους για αυτή τη συζήτηση. Είχαμε τις διαφορετικές κατηγορίες, τους διαχωρισμούς, τις διαφορετικές έννοιες, ε, διακρύβωση όλων αυτών, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή ανάλυση. Είχαμε παρουσίαση πολλών και διαφορετικών καταστάσεων και έτσι μπορέσαμε να αντιληφθούμε καλύτερα τι είναι αυτή η μάχη, αυτός ο αγώνας ε, κατά πολέμησης της εμπορίας ανθρωπίνων όντων. Ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντες, όλους τους ομιλητές, τις ομιλήτριες, τους συναδέλφους και τις συνεδέλφους που είναι εδώ παρόντες και παρούσες. Ολοκληρώνεται αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας και θα έχουμε μια, ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών, τριών λεπτών, για να ξεκινήσουμε το επόμενο κομμάτι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

Okay.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 Voilà, on va commencer. Merci. Ah, c'est beau ça. Voilà, merci à tout le monde. Λοιπόν, ε, θα, ξανα... θα συνεχίσουμε τώρα. Διήρκησε ήδη υπερβολικά το διάλειμμα αυτό. Πέντε λεπτά ολόκληρα. Δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας. Ε, σήμερα ε, έχει οργανωθεί αυτή η συζήτηση ε, για τις σχέση μας με τη Λευκορωσία και έχω την χαρά εξάλλου να έχω δίπλα μου τον συνάδελφο Ζωεύσκη που είναι ε, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Οι συζητήσεις μας είναι ε, σημαντικές γιατί το πολιτικό τοπίο της χώρας αλλάζει και γίνονται επίσης ε, σημαντικές αλλαγές στην ε, γειτονιά μας. Σύντομα, εξάλλου, θα έχουμε τη διάσκεψη κορυφής στη Ρήγα, 21 και 22 ε, Μαΐου. Ε, εν τω μεταξύ, η Λευκορωσία θα πρέπει να παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και χαίρομαι που σήμερα έχουμε προσώπους που θα μιλήσουν για την κατάσταση στη χώρα αυτή. Ε, είναι σαφείς ε, οι θέσεις μας ε, ε, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ε, κρατάει μια στεναρή στάση απέναντι στη Λευκορωσία σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν πέρυσι. Μέχρι τον... και πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τον Οκτώβριο φέτος. Και θα πρέπει να συνεχίσει επίσης τη συνεργασία που θα αποσκοπεί, θα αφορά κυρίως την κοινωνία των πολιτών και τα τεχνικά ζητήματα. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάθε βελτίωση των διμερών σχέσεων θα πρέπει να εξαρτάται από μια σημαντική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη χώρα. η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω η Κομισιόν ε, διεξάγουν συζητήσεις όσον αφορά τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Ε, στις 12 Μαρτίου ε, έγινε η σχετική, ελήφθη η σχετική απόφαση. Το Κοινοβούλιο ε, ε, βλέπει θετικά την εξέλιξη αυτή, αλλά το πραγματικό τεστ της δημοκρατίας ε, θα είναι οι επόμενες προεδρικές εκλογές το Νοέμβριο του 2015. Θα πρόκειται για μια πραγματική δοκιμασία, ένα πραγματικό τεστ. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ε, προηγουμένως όμως επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο τον συνάδελφό μου, τον πρόεδρο της ε, αντιπροσωπείας μας για τις σχέσεις με την ε, ε, Λευκορωσία, τον κύριο Ντροζιεύσκη. Bardzo serdecznie przywitać i też Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι έχουμε εδώ τον Άλες Μπιαλιάτσκι. Σας καλωσορίζω μπορέσατε να αποφυλακιστείτε επιτέλους και μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα. Ε, καλωσορίζω και τους καλεσμένους μας από την Μόσχα, οι οποίοι αναλύουν την κατάσταση στη Λευκορωσία ε, με διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με αυτή που υιοθετούν οι Βρυξέλλες. Ωστόσο η συνεισφορά σας στη συζήτηση είναι πολύτιμη και σας ευχαριστώ θέρμα. Κυρίες και κύριοι, δέχτηκα αυτή την πρόταση διοργάνωσης κοινή συνεδρίασης, γιατί η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά σημαντική για τη Λευκορωσία. Το ενδιαφέρον ε, για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα αυτή εντάθηκε λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε η Λευκορωσία ως διαμεσολαβητής στην σύγκρουση της Ουκρανίας μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σχολιάζοντας όλα αυτά, ωστόσο ο χρόνος δεν υπάρχει. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω δύο-τρία στοιχεία. Οι τελευταίες εκλογές στη Λευκορωσία χαρακτηρίστηκαν μη δημοκρατικές, δεν εκπλήρωσαν τα διεθνή πρότυπα για τη δημοκρατικότητα των εκλογών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημες σχέσεις με το ε, Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας ως εκ τούτου και γι' αυτό το λόγο μεταξύ άλλων δεν προσεκλήθη το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας να συμμετάσχει στο Euronest κοινοβουλευτική, διακοινοβουλευτική συνάντηση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας και ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας. Και τα τρία βασικά ζητήματα είναι τα εξής. Υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία. Συνεχίζουν, συνεχίζουν να υπάρχουν και πρέπει να είναι σημαντικό ζήτημα σε αυτή την ε, επικοινωνία. Άλλο πρόβλημα είναι η χρήση της ε, θανατικής ποινής, η οποία ισχύει στη Λευκορωσία και έχει εφαρμοστεί και φέτος μάλιστα, όχι μόνο τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής τουλάχιστον. Και τρίτο πρόβλημα είναι η ελευθερία του τύπου. Ε, σε σχέση με τις τελευταίες αλλαγές ε, στη σχετική νομοθεσία της χώρας αυτής. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά η έκφραση καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών ε, ενδιαφερόντων, ο σεβασμός στη γλώσσα της Λευκορωσίας, όλα αυτά θα πρέπει να τηρούνται και να γίνονται αντικείμενο σεβασμού, να μπορεί κανείς να εκφραστεί καλλιτεχνικά και στη γλώσσα της Λευκορωσίας μεταξύ άλλων. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά όλα αυτά ε, πρέπει να ενταθούν, να εφαρμοστούν. Έχουμε μια σειρά συμφωνιών, πλησιάζουμε σε αυτές μάλλον για οικονομική στήριξη και θα πρέπει η οικονομική στήριξη να δίδεται έχοντας εγγυήσει ότι μπορούν να ακουστούν και άνθρωποι που ε, σκέφτονται ε, διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρώτο μας προσκεκλημένο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς και για μεγάλη μας χαρά που μπορούμε να σας υποδεχθούμε εδώ. Κύριε Άλες Μπιαλιάτσκι, είστε πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βιάσνα, το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν πριν από 20 χρόνια, το 1996. Όπως θα γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μπιαλιάτσκι είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα γνωρίζετε κυρίες και κύριοι επίσης ότι ο κύριος Μπιαλιάτσκι πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή, απελευθερώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και η δίκη του έτυχε γενικότερης καταδίκης από τη διεθνή κοινότητα. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλημμένως έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας, έχουμε ζητήσει την απελευθέρωσή του. Για Πολλά χρόνια ο κύριος Μπιαλιάτσκι ήταν ακτιβιστής ε, και προσπαθούσε να αγωνιστεί ενάντια των φρικτών απολυταρχικών καθεστώτων που υπήρχαν στη χώρα αυτή. Έρχεται σήμερα να ε, μας μιλήσει για την εμπειρία του. Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βιάσνα είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι διαδίδει πάρα πολλά στοιχεία και πληροφορίες για την καταστρατήγηση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα ο κύριος Χάν είναι στο Μίνσκο, ο αρμόδιος επίτροπος για τις ε, σχέσεις ε, γειτονίας. Ο επίτροπος Χάν είναι στο Μίνσκ σήμερα και ο κύριος Μπιαλιάτσκι είναι εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, υπάρχει λοιπόν διερμηνία από τα ρωσικά στο κανάλι 24. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που δίνει ε, σε ακτιβιστές για πολιτικά και ατομικά δικαιώματα στην Λευκορωσία και για όλους αυτούς που ήταν θυμάτα καταστολής τα τελευταία χρόνια το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, μιλάει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναφέρεται και στο όνομά μου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι διώξεις αυτές ε, που λαμβάνουν χώρα στη Λευκορωσία. Και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και επίσης να πω την τελευταία φορά που μίλησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ε, τον Ιούλιο του 2011. Δύο εβδομάδες αργότερα βρέθηκα στη φυλακή. Ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί ε, αυτό το προηγούμενο σενάριο και αυτή τη φορά. Η ομιλία μου εκείνη την φορά ήταν αφιερωμένη στην ε, κατάσταση όσον αφορά τις εκλογές ε, του 2010. Η κατάσταση ήταν όντως κρίσιμη. Ε, σας υπενθυμίζω ότι 50 άτομα φυλακίστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εκλογές το 2010. Κάποιοι από αυτούς υποψήφοι για πρόεδρος, για τη θέση του πρόεδρου. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετεί μια πολύ σκληρή ε, στάση απέναντι στην Λευκορωσία. Ε, ζητάει ε, κυρώσεις για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο γιατί τον Αύγουστο του 2012 40 άτομα απελευθερώθηκαν, πήραν αμνηστία. Πιστεύω ότι το πακέτο των κυρώσεων που υιοθετήθηκε το 2011 ε, παραμένει πάντα επίκαιρο ε, μέχρι ότου να μην υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στην ε, Λευκορωσία. Ένας από τους προεδρικούς υποψηφίους του 2010 βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Φέτος τον Νοέμβριο θα έχουμε και πάλι οι προεδρικές εκλογές και μια εκλογική διαδικασία. Το όλο όμως θέμα το έχουν στα χέρια τους και πάλι οι αρχές της Λευκορωσίας. Δεν υπάρχει λοιπόν από ό,τι βλέπω κανένας λόγος να εγκατελειφθούν οι κυρώσεις για το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Η κατάσταση ε, είναι ότι ε, όπως είπατε ε, αποφυλακίστηκα πριν από 11 μήνες έχω αναλάβει τις δραστηριότητές μου ταξιδεύω παντού αλλά πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς τους μήνες αυτούς δεν διαπίστωσα καμία βελτίωση αφότου αποφυλακίστηκα. Μπορεί με μονομένες περιπτώσεις να υπάρχουν, αλλά γενικά η κατάσταση είναι εξίσου θλιβερή όπως και στο παρελθόν. Ε, αντίθετα μπορούμε να δούμε κάποια σημάδια επιδείνωσης της κατάστασης που σχετίζονται και πάλι με την προεκλογική ε, αυτή περίοδο εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Βλέπουμε ότι οι αρχές της Λευκορωσίας φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο ε, της κατάστασης παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς ε, η νομοθεσία σχετικά με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ε, έγινε ακόμα πιο σκληρή. Ε, οι αρχές έκλεισαν ανεξάρτητα websites, ανεξάρτητες ιστοσελίδες ε, με νομοθεσία η οποία είναι αντίγραφο της ε, ρωσικής νομοθεσίας. Ε, βλέπουμε την άμεση επιρροή του ανατολικού μας γείτονα σε σχέση με τον τρόπο ελέγχου των πληροφοριών, της ενημέρωσης υπάρχουν ε, ε, διαδικασίες στα ε, διοικητικά δικαστήρια που στρέφονται εναντίον των ανεξάρτητων δημοσιογράφων που εργάζονται στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν τέτοιες δίκες, υπάρχουν έρευνες κατοίκων, κατάσχονται υπολογιστές ε, και οι αρχές της Λευκορωσίας χρησιμοποιούν τα μέτρα αυτά για να περιορίσουν την ροή των πληροφοριών και να εμποδίσουν τη δουλειά των ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Ε, το εύρος η κλίμακα ε, των μέτρων αυτών αυξάνεται συνεχώς. Ε, η κυβέρνηση εισάγει ε, νέα νομοθεσία για τη φορολόγηση των ανέργων. αυτό σημαίνει ότι κάθε άνεργος θα πρέπει να πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό για την κοινωνική πρόνοια. Δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά, γιατί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας αποτελείται από άτομα που έχουν απολυθεί από τη δουλειά τους. Ε, πρόκειται για τα πιο ευάλωτα άτομα της κοινωνίας. Το εκλαμβάνουμε αυτό ως ε, ένα συγκεκριμένο πολιτικό ε, δείγμα προσπάθειας ελέγχου της κοινωνίας. Οι αρχές θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία και επίσης να πιέσουν, για να πιέσουν οι αρχές τους ανθρώπους ε, να ε, δουλέψουν. Παρόλο που το Συνδέμα μιλάει για την εργασία ως δικαίωμα. Φαίνεται όμως ότι η εργασία ε, τίνει να γίνει καταναγκαστική εργασία. Θα θυμάστε ότι ο Τζόσεφ Πρόσκι ε, φυλακίστηκε διότι δεν δούλευε θεωρήθηκε ότι ήταν κυφίνα. Νομίζω ότι έχουμε μια παρόμοια κατάσταση στην ε, Λευκορωσία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα ε, που ε, δείχνει ότι στην Λευκορωσία επαναλαμβάνονται πράγματα που έγιναν στη Ρωσία πριν από 20 και 25 χρόνια. Παράλληλα προσπαθούμε να αποφύγουμε μια οικονομική κρίση που φαίνεται να απειλεί τη χώρα. Πέρυσι ε, κατέρευσε η ισοτιμία, το ρούβλι της ε, Λευκορωσίας έχασε 40% της αξίας του και σχεδόν όλοι οι Λευκορώσοι έγιναν φτωχότεροι κατά 40% και ο, ο, ο κίνδυνος της οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο σοβαρός. Ε, αντίθετα όμως με αυτή την ζωφερή εικόνα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια αισιόδοξη ε, αφήγηση όσον αφορά ε, τις σχέσεις ε, της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ίσως και γίνεται λόγος για βελτιωμένες ε, ε, σχέσεις, πράγμα το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα πραγματικά ε, συμβαίνουν στη χώρα. Είναι σαφές ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έλαβε εντολές να βελτιώσει πάση θυσία τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των περχόμενων εκλογών, ώστε η εικόνα να απαλληθεί κάπως και επίσης ε, ε, προσπαθούν να αποφύγουν ε, το οικονομικό κράχ. Δεδομένου ότι η, σχέσεις, η βοήθεια μάλλον από τη Ρωσία ε, φθήνει και γι' αυτό ο Λουκασέγκο ψάχνει νέες πηγές χρηματοδότησης. Το θέμα είναι ε, να μην ε, βοηθηθεί το καθεστώς ε, με τη διαδικασία αυτή εις βάρος των, της κοινωνίας των πολιτών. Διότι σας λέω ότι παρόλε τις αλλαγές που ενδεχομένως συμβαίνουν στη Λευκορωσία, τα χρήματα θα χρησιμεύσουν για την υποστήριξη του καθεστώτος. Όσον αφορά τον Λουκασέγκο, ε, υποστηρίζοντας τον Λουκασέκο, στην πραγματικότητα ε, υποστηρίζουμε τον Πούτιν, γιατί είναι οι, πάρα πολύ στενοί συνεργάτες. Υπάρχει πολιτική, στρατιωτική, οικονομική συνεργασία σε μαζική κλίμακα. Πολύ πρόσφατα ε, υπήρξαν συμμαχίες ε, που ε, συμμετείχαν και η Ρωσία και η ε, Λευκορωσία, διάφορες μορφές ε, συνεργασίας, βρασιατική συνεργασία κλπ. που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αντίβαρο ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να πιστεύουμε τα λόγια της, ε, του καθεστώτος της Λευκορωσίας, να δούμε μόνο ε, τις πράξεις τους. Ε, έχουν ενταθεί επαφές τους τελευταίους μήνες. Οι επαφές αυτές όμως θα πρέπει να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Διότι διαφορετικά οι επαφές αυτές θα χρησιμεύσουν μόνο για να υποστηρίξουν το καθεστώς. Ε, να στηρίξουν το καθεστώς χωρίς την ουσία να αλλάζουν τίποτα στη δομή της ε, κοινωνίας της Λευκορωσίας. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών ε, της Λευκορωσίας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτή και θεωρούμε ότι η ενίσχυση των διπλωματικών επαφών ε, και οι επαφές με τους διπλωμάτες στο Μίνσκ ε, δεν θεωρούμε ότι θα επηρεάσουν κατά κανένα τρόπο κατά, κατά κανένα σημαντικό τρόπο ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Επίσης το θέμα των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό. θεώρηση θα γίνει φτηνότερη, η βίζα θα γίνει φτηνότερη και ίσως στο μέλλον να, ε, ε, να μην χρειάζεται και η Λευκορωσία ε, βίζα, όπως και η Μολδαβία και η Ουκρανία ενδεχομένως. Και αυτό ίσως θα είναι το πιο χρήσιμο μέτρο από ότι όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μαζί. Ευχαριστώ. Euh, bienvenue également. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μίκλος Χαραστή, ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Ασκεί τα καθήκοντα αυτά εδώ και δύο χρόνια περίπου, ενώ πριν ήταν εκπρόσωπος για την ελευθερία των μέσων επικοινωνίας του ίδιου οργανισμού έχει συμμετάσχει ως παρατηρητής σε ε, πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στο Τατζικιστάν για παράδειγμα ήσασταν. Και παρακολουθεί την κατάσταση στη Λευκορωσία σε διαβούλευση με διαφόρους εταίρους, ενώ η πρόσβαση στη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τις εκθέσεις του ε, για το θέμα αυτό. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι μπορώ να μιλήσω μετά τον κύριο Μπιαλιάτσκι. Και χαίρομαι διότι αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον εκείνος έχει ελευθερωθεί. Είναι όμως ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή μπορεί να ταξιδέψει μέχρι εδώ. Τίθεται το ερώτημα. Ας ε, θέσουμε το θέμα των πολιτικών κρατουμένων στην ευρύτερη του έννοια. Τι σημαίνει να ελευθερώνεται κάποιος επειδή ο κάθε πρόεδρος δίνει αμνηστία ή επειδή ολοκληρώνεται ε, τα χρόνια κατά την ε, οποία ε, έπρεπε να εκτίσει την ποινή του. Συγγνώμη, θέλετε να βγάλω το, τη διαπίστευσή μου για τη φωτογραφία. Εντάξει. Ό,τι πείτε. Δεν έχω πρόβλημα. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, μπορεί να ελευθερώνεται ε, αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία στην οποία αναφέρθηκε ο Άλες Μπιαλιάτσκι, ότι δηλαδή θεωρούνται παράσιτα ή ότι είναι στο περιθώριο. Δεν έχει νόημα να ελευθερώνεται κανείς εάν δεν αποκαθίσταται ε, το καθεστώς του, η ιδιότητά του, αν δεν αποκαθίσταται η αλήθεια για το πρόσωπό του. Ή αλλιώς έχουμε αυτόν τον αντικατοπτρισμό ότι η αλλιώ έχουμε αυτό τον αντικατοπτρισμό, τάχα η ψευδέστηση ότι τάχα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Οφείλω να σας πω και πολύ σύντομα θα το υποβάλω και στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εδρεύει στη Γενέβη και αποτελεί μέρο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οφείλω να σας πω λοιπόν ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά έχει και υποβαθμιστεί λόγω των κανονισμών, των κανονιστικών διατάξεων, των δυνατοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, της, λόγω της υποβάθμισης της ανθρώπινης ζωής ε, στην χώρα αυτή, στη Λευκορωσία. Και μάλιστα η κατάσταση με τα ελευθερία του τύπου έχει επιδεινωθεί είναι τα τελευταία 20 χρόνια ένα εργαστήριο όπου γεννιόνται νέα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια η χώρα αυτή. Είναι ένα εργαστήριο όπου ε, υψώνονται διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για να αποκτήσει το κράτος πάλι έλεγχο του χώρου ε, της ελευθερίας του τύπου, του διαδικτύου μεταξύ άλλων και τα καταφέρνει κιόλα. Ε, υπάρχει μεγάλο πλήγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε, του οτιδήποτε μπασχεπτώσει λαμβάνει η χώρα στη δημόσια σφαίρα. Στη Λευκορωσία κάθε μέρα η έννοια του τι είναι δημόσια δραστηριότητα, τι είναι δημόσια δράση, τι είναι δημόσια παρουσία στους δρόμους, τιμωρείται όλο και περισσότερο εάν λαμβάνει χώρα χωρίς άδεια. Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει καθόλου είναι η λαμπρή εφεύρεση της Λευκορωσίας για την τριπλή παγίδα οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας. Είναι συνέρχεστε, είναι συνεταιρίζεστε, είναι μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οποιαδήποτε δραστηριότητα και να θέλει κανείς χρειάζεται άδεια για να την κάνει. Καμία σχεδόν δεν εγκρίνεται η άδεια για καμία σχεδόν από τις αρχές. Και η τρίτη παγίδα είναι ότι είναι ποινικό κολάσιμο και διώξιμο, όχι μόνο να οργανώσει κανείς κάτι για το οποίο δεν έχει πάρει άδεια, αλλά είναι ποινικό κολάσιμο και διώκεται να συμμετάσχει πολύ απλά σε αυτό. Άρα ο κύριος Μπιαλιάτσικη έχει ελευθερωθεί, έχει αποφυλακιστεί, είναι εκτός φυλακής λόγω της επιοίκειας του Προέδρου, διότι το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διάσνα του οποίου προεδρεύου είναι μια εξαιρετικά σημαντική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πήρε την καταχώρηση και άρα από τη στιγμή που ηγείται αυτή τη οργάνωση είναι εγκληματία. Δηλαδή, ο κύριος Μπιαλιάτσκι είναι σήμερα μαζί μας γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ακόμα εκδώσει την εντολή να ξαναφυλακιστεί επειδή είναι πρόεδρος μιας οργάνωσης της Βιάσνα η οποία δεν πήρε πάλι άδεια λειτουργίας. Επομένως, βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ο πρόεδρος τα 20 τελευταία χρόνια είναι ο απόλυτος ηγέτης της χώρας. Ε, κατ' ουσίαν, ονομαστικά αν θέλετε, η Λευκορωσία έχει κοινοβούλιο, η χώρα όμως κυβερνιέται με προεδρικά διατάγματα. Δύο είναι τα είδη της δικαιοδοσίας του Προέδρου. Ε, το ένα δίδεται από το Σύνταγμα και το δεύτερο από τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου. Και αυτού του είδους η δικαιοδοσία και η νομολογία καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Δεν υπάρχει διαφυγή. Είναι το μόνο κοινοβούλιο στην Ευρώπη το οποίο τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει κανενός είδους αντιπολίτευση. Είναι ένα κοινοβούλιο που δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και συν της άλλης, κάθε φορά που εκλέγεται ο πρόεδρος είναι μαζική η εκδήλωση της βίας στους δρόμους. Επομένως, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ούτε σε πολιτικό επίπεδο ούτε σε κοινωνικό επίπεδο, παρόλο που Υπάρχει ο μύθος ότι η τάχα είναι ε, κράτος πρόνοιας η Λευκορωσία. Σε καμία περίπτωση. Ε, είναι μια κοινωνία όπου είναι μια οικονομία με ε, καταναγκαστική εργασία σε μεγάλο βαθμό. Το 70-80% των επιχειρήσεων ανήκουν στο κράτος και όλοι εμείς που έχουμε ζήσει ε, στο κομμουνιστικό καθεστώς θυμόμαστε αυτή τη ψευδή ασφάλεια, τη ψευδή ε, σταθερότητα που δίδει ως εντύπωση ένα κράτος στους ε, πολίτες όταν οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην ιδιοκτησία του. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι πάρα πολύ αδύναμα στη Λευκορωσία, όλα εξαρτώνται, ενώ τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ ευπαθή και όλα εξαρτώνται από την εξουσία του Προέδρου. Ε, πιστεύω ότι εάν έτσι έχει η κατάσταση και λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης έχει υπάρξει ενδεχομένως ή έχετε δει εσείς βελτίωση ε, της κατάστασης της Λευκορωσίας διότι έγινε χώρα διαμεσολαβήτρια στην κρίση στην Ουκρανία Εάν το αντιλαμβάνεστε έτσι τα πράγματα, αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσετε ως πρόβλημα είναι το εξής. Ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρχει μια δίτη πολιτική εναντί της Λευκορωσίας. Δηλαδή από τη μία ε, πλευρά να επιδεινώνεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπάρχει αυτός ο παράγοντας που να επιδεινώνει το κλίμα, η πολιτική ε, κρατούμενοι υπάρχουν, τα νούμερα τους άλλοτε να αυξάνονται, άλλοτε να μειώνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση να συνεχίζουν να υπάρχουν και το σύστημα κανονιστικών διατάξεων να μην αλλάζει και η δημοκρατία και ο πλουραλισμός να μην βελτιώνονται, αυτό από τη μία και από την άλλη θα έχετε ε, θερμή διπλωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση των σχέσεων και της κατάστασης με την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμβάλλει. για να συγκεράσει, ε, να κάνει να πλησιάσει το ένα το άλλο αυτά τα δύο διαφορετικά πεδία που μόλις τώρα ανέφερα. Η αιρεσιμότητα, αυτό το οποίο ανέφερε ο πρόεδρος, το conditionality δηλαδή, θα πρέπει να είναι κάτι που να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να έχουμε βαθμιά προσέγγιση, τίποτα δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα, δεν μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα σε μια στιγμή μέτρο όμως της βαθμιαίας ε, προσέγγισης θα πρέπει να εφαρμοστεί και να υιοθετηθεί στις σχέσεις με την Λευκορωσία. Δηλαδή αυτά που δανείζουμε ουσιαστικά ε, θα είναι στήριξη στην πολύ κατασταλτική έννοια της σταθερότητας και της ασφάλειας του καθεστώτος. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος τελικά να δανείσουμε και αυτό έτσι να ερμηνευθεί και έτσι να μεταφραστεί και τελικά να προσυπογράψουμε στις καθημερινές προειδοποιήσεις του Προέδρου Λουκασένκο ότι δηλαδή αντιτιθέμεθα στις προσαρτήσεις δεν μας, δεν μας αρέσει η παραβίαση της εδαφικής ακαιρεότητας από την άλλη πλευρά όχι πλατεία Μαϊντάν. Και αν μεταφράσει κανείς την προειδοποίηση όχι Μαϊντάν με όρους αλήθειας, τότε βλέπει ένα πολύ κατασταλτικό και πολύ καλά σχεδιασμένο σύστημα καταπίεσης όπου δεν μπορούν ε, οι πολίτες να ασκήσουν τα ανθρώπινα και δημοκρατικά τους δικαιώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι Πρέπει το Κοινοβούλιο να ε, αξιοποιήσει ε, κάθε δυνατή καινοτομία, εφευρετικότητα και επινοητικότητα που έχει έτσι ώστε να συνδέσει τη βαθμία προσέγγιση με τη Λευκορωσία ε, με την απέτηση για βαθμία βελτίωση των, της κατάστασης επιβάλλοντας όρους και προϋποθέσεις Όπως και ο Άλες αναφέρθηκε, ο Άλες Μπιαλιάτσκι, το σύστημα του Προέδρου Λουκασένκο χρειάζεται την Ευρώπη πραγματικά σήμερα. Και παρόλο που η Λευκορωσία έχει γίνει μέλος της Ευρασιατικής Ένωσης και παρόλο που υπάρχει αυτή η Ευρωασιατική Ένωση, η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκονται οι χώρες αυτές και κυρίως η Ρωσία δείχνει ότι θα είναι δύσκολο να συνεχιστούν ε, οι να παραμείνουν ανοιχτές οι παραδοσιακές οδοί στήριξης στη ε, Λευκορωσία, αυτές που ε, κάνουν το σύστημα Λουκασένκο να συνεχίσει να ε, υπάρχει και να επιβιώνει. Άρα η Λευκορωσία χρειάζεται την Ευρώπη και θα πρέπει η βοήθεια της Ευρώπης να εξαρτάται από, την, από όρους και προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια προσωπική παρατηρήση. Ξέρετε, οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν θα αναγνωρίσουν την εντολή αυτή. Εγώ πιστεύω ότι είναι συμβολικό το ζήτημα που σημαίνει, που αποκαλύπτει, που λέει πολλά για την ικανότητα και τη βούληση ε, του συστήματος να συνεργαστεί με την διεθνή τάξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, για να είμαι πιο αποτελεσματικός. Ελπίζω από ότι ε, είμαι σήμερα, χρειάζομαι βίζα. Πρέπει να μπορώ να μπω στην επικράτεια της Λευκορωσίας, να μου επιτραπεί και λένε ότι δεν αναγνωρίζουν την εντολή μου εξού και δεν μου εκδίδουν. Όμως, για να πάρουν σοβαρά το Διεθνές Σύστημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, για να πάρουν σοβαρά την ανάγκη να συνεργαστούν με εσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να του πείτε ότι η εντολή αυτή την οποία διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων στις συναντήσεις της Γενέβης ισχύει και απαιτεί τη συνεργασία της Λευκορωσίας. Πρέπει να στείλετε επιγόντως αυτό το μήνυμα και θα σας είμαι ευγνώμων αν μπορείτε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στο Μίνσκ. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, στον κύριο Αντριάνο Μάρτινς, ε, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ε, σκοπεύει να παραμείνει εμπλεγμένη στην Λευκορωσία και στον πολυμερή διάλογο για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντο, καθώ και να συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία των πολιτών και γενικά τον λαό τη Λευκορωσίας. Ταυτόχρονα, με δεδομένη τη σοβαρή ανησυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, τον Οκτώβριο του 2014 το Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση για άλλο ένα έτος των περιοριστικών μέτρων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους ε, είδαμε πιο θετικές ε, τάσεις στην συμπεριφορά της Λευκορωσίας απέναντι στην Δύση. Μια πιο μια διαφορετική στάση με περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα ή δυνατότητα να φιλοξενηθεί ένας ε, διμερής διάλογος, διαπραγματεύσεις βίζας και επανεισδοχής, ε, καθώς επίσης και η αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων με την Σουηδία, την απελευθέρωση του Άλες και πολιτικού κρατούμενου, διοργάνωση διαφόρων σεμιναρίων από κοινού με την κοινωνία των πολιτών και ενεργό συμμετοχή στην ενδιάμεση φάση ζητημάτων εξυγχρονισμού. Το περιφερειακό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε έχει αλλάξει. Η Λευκορωσία λοιπόν δεν ακολούθησε την πορεία που περίμεναν πολλοί, ότι δηλαδή θα ακολουθεί το κάθε βήμα της ε, Ρωσίας. Αντιθέτως, έχει κάνει μια σειρά θαραλέων βημάτων ε, και στο θέμα της Ουκρανίας και της εκεί σύγκρουσης, παραδείγματος χάρη όταν η Ρωσία ακύρωσε τις εισαγωγές ε, κρασιού από τη Μολδαβία αύξησε τις εισαγωγές της η Λευκορωσία. Για να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το παράθυρο ευκαιρία, τα κράτη-μέλη τον Ιανουάριο έκαναν έναν κατάλογο 29 μέτρων για να εμβαθύνουν την ε, πολιτική μιας ε, κριτικής έμπλοκης με την Λευκορωσία. Έτσι λοιπόν είχαμε την ε, συνάντηση της ε, Χέλγα Σμίτ Γενικής Γραμματέως ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με τον πρόεδρο Λουκασένκα το Μάρτιο. Όμως, παρά τις πιο θετικές τάσεις στις σχέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί να κάνει περαιτέρω βήματα λόγω μόνο του θετικού ρόλου της Λευκορωσίας στην Ουκρανία. Και αυτό το είπαμε στον πρόεδρο Λούκασέγκο στην επίσκεψη του Μαρτίου. Του είπαμε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και δεν θα ξεχάσει τις ανησυχίες της που αφορούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει μόνο μικρά και ιστοριακά βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων της με την Λευκορωσία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Κύριε Οστρεβίσιος, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Άλεξ Βιαλάτσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάδελφοι, θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο θαραλέο είναι εκ μέρους του το να επισκέφτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μια τυχαία επίσκεψη. Ε, δεν έχει καμία εγγύηση. Από τη στιγμή που θα επιστρέψει στο Μίνσκι θα περάσει τα σύνορα της Λευκορωσίας ότι δεν θα ε, που θα καταλήξει καθώς θα προέρχεται από τη Δύση. Και αυτό είναι ε, ένα λαμπρό παράδειγμα της ελεύθερης βούλησης ενός ανθρώπου που ε, θέλει ένα διαφορετικό μέλλον και έχει μια διαφορετική κατανόηση ε, της Λευκορωσίας ως έθνους και ως χώρας. Θα πρέπει πραγματικά να τον συγχαρούμε και να του ευχηθούμε να συνεχίσει να είναι αφοσιωμένο σε αυτό το σκοπό. Βλέπουμε μια δεν βλέπουμε καμία αλλαγή πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Λευκορωσία. Δεν βλέπω ε, καμία θετική κίνηση του Λουκασάνικου απέναντι στη Δύση. Δεν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι σχετικά με αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή ο Λουκασάνικο, γιατί ε, βρίσκεται εν ώψη εκλογών και είναι ένας πολύ έξυπνος πολιτικός. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πριν από τις εκλογές, λοιπόν, πριν από ε, κάποια σημαντικά γεγονότα, αλλάζει την πολιτική του και λόγω αυτού ε, υποφελείται σε πολύ σημαντικό βαθμό, όπως έγινε και πριν από τις εκλογές του 2010. Η ε, ε, επανεκλογή, μάλλον θα πρέπει να πούμε, είναι αυτό που θα συμβεί φέτος και όχι οι εκλογές. Είναι πιο ακριβής όρος. Ε, δεν θα συμφωνήσω με την ε, ε, αισιόδοξη στάση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία ψήφισε μαζί με τη Ρωσία κατά της Κρυμαίας και αυτό είναι εντελώ απαράδεκτο. Η Λευκορωσία είναι μέλος της κοινοπολιτείας δηλαδή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Ε, ο Πούτιν και πάλι σε κάθε ευκαιρία ε, κατακρίνει τη Δύση, σε κάθε συνέντευξη που δίνει. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τον Άλεξ, μια που έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η αποφυλάκηση πολιτικών κρατουμένων και η αποκατάστασή τους είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα. Γιατί ένα πράγμα είναι ο Λουκασέγκο να απελευθερώσει ένα πολιτικό κρατούμενο και εντελώ διαφορετικό να τον αποκαταστήσει ε, στην κοινωνία. Ε, το βάρος... Ε, ε θα τον βαραίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη ζωή του. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι απαιτήσει θα πρέπει να θέσει η Δύση πριν από τη Σύνοδο Κορυφή στη Ρήγα. Ε, γιατί κάτω τους προσεχείς μήνες ε, θα πρέπει να δούμε ε, με πολύ προσοχή τι θα γίνει. Ο Λουκασέγκο μπορεί να κληθεί, να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής στη Ρήγα. Είναι πιθανόν ε, οι Ευρωπαίοι ηγέτε λοιπόν και ο Λουκασέγκο να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλες τις πολιτικές μας και όλες τις αξίες και τις αρχές μας. Τι απαιτήσει λοιπόν θα πρέπει να έχουμε σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, υιοθετεί μια πολύ αυστηρή πολιτική γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής ε, στη Ρήγα, αν πρόκειται να προσκληθεί ο Λουκασέγκο. Θα πρέπει να είμαστε αφήσει τι θα πρέπει να κάνει ο Λουκασέγκο έως τότε. Ευχαριστώ. ομιλητής. ευχαριστώ. Χαιρετίζω και εγώ τον κύριο Μπιαλιάτσκι Καταλαβαίνω και την ψυχή του κατάσταση, λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά που πέρασε και την αβεβαιότητά του για το μέλλον. Ε, τον ευχαριστούμε λοιπόν που βρίσκεται εδώ και προσπαθούμε με τη βοήθειά του να καταλάβουμε τι είναι δυνατόν να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ακούσει περισσότερο η φωνή του στο ΜΙΝΚ και προς τον Λουκασέγκο. Εξάλλου, όπως είπατε και εσείς, η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Υπάρχει μια επιδείνωση ανευπροηγουμένου όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα. Και αυτό το έχουν καταγγείλει πολλοί. Πολύ πρόσφατα ο Λουκασέγκο ε, ε, φιλοξένησε ε, την Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία και αυτό ε, έδωσε μια λάμψη στην εικόνα του. αλλά θα ήθελα να να κάνω ορισμένε ερωτήσεις. Ε, προηγουμένως όμως μια παρατήρηση ε, για αυτά που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ γενικά ε, βλέπω με κάποια δόση real politik της διεθνή μας σχέσης. Το να κάνουμε όμως μικρά τέτοια βήματα απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση ε, δεν είναι η σωστή απάντηση πιστεύω ότι πρέπει να ενεργήσουμε σε δύο άξονες κατά κύριο λόγο. Πρώτον, θα πρέπει παρόλο τις δυσκολίες που έχει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΜΙΝΣ, να κάνουμε ε, σαφές ότι θα πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, παρόλο που αυτό αποτελεί ε, μέρος της νέας ε, διαδικασίας που αποφασίσαμε στο που υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που περιλαμβάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιό της. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το πρόβλημα και να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε σκόπιμο και χρήσιμο να τοποθετηθεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ε, αν θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό θα μπορέσει να ασκήσει κάποια πίεση, μια τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να αλλάξει στο άμεσο μέλλον η πολιτική που ε, ασκεί ο Λουκασέγκο. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνακ. Well, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω πως ε, στην πρώτη μου θητεία το 2003 με ρώτησαν για την ε, Λευκορωσία και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα χειροτέρευσαν τα πράγματα. Είχα δώσει μία συνέντευξη σε μία πολωνική εφημερίδα και έλεγα πως ε, η Λευκορωσία ήταν η Κούβα της Ευρώπης η οποία ε, η Κούβα εντωμεταξύ η ίδια έχει αρχίσει να ανοίγει στον έξω κόσμο, αλλά η Λευκορωσία έχει μείνει κολλημένη σε αυτή την κατάσταση μονοκομματικής, αυταρχικής διακυβέρνησης, ε, ε, μια δικτατορία τύπου χώμο Σοβιετικούς με μια κάγκεμπέ που λειτουργεί ακόμα. Με καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κάποια ελεύθερη αγορά λίγο κινείται η οικονομία και έτσι η μεσαία τάξη και η νομεκλατούρα μπορεί να απολαμβάνει κάποια προνόμια της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης αλλά είναι πολύ περίεργη η κατάσταση είχα πάει πριν από λίγα χρόνια και δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει πολύ Τώρα ίσως υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας δεδομένης της ανόδου του πουτινισμού και της επιθετικής επέκτασης της Ρωσίας με την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας ε, και αυτού του πολέμου στην ε, Ουκρανία. Ίσως ο Λουκασένκο έχει αρχίσει να ανησυχεί για το ποια είναι τα σχέδια του Πούτιν. Πριν από καμιά δεκαετία ο Λουκασένκου με την ένωση με την Ρωσία ε, νόμιζε ότι κάποια στιγμή θα βρισκόταν ο ίδιος στο Κρεμλίνο ως ηγέτης των δύο ηγετών. Αλλά ε, από ό,τι φαίνεται ο Πούτιν απλά σκοπεύει να καταστήσει την Λευκορωσία μια περιφέρεια της Ρωσίας. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επαφές, αλλά οπωσδήποτε τα 16 χρόνια που είμαι εδώ ε, Ευρωβουλευτή για ζητήματα εξωτερικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Επαφές, μη επαφές, στοχευμένε κυρώσει, Τίποτα δεν αλλάζει την κατάσταση. Ίσως να ξαναπροσπαθήσουμε τώρα δεδομένης ε, της γεωπολιτικής ε, αλλαγής ε, στην ε, Ρωσία του Πούτιν αλλά θα πρέπει να έχουμε σχέσεις ε, με την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας έχω συναντήσει πάρα πολλούς αντιφρονούντες και ηγέτες της αντιπολίτευσης και οπωσδήποτε η ομάδα μου το ECR η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του Κοινοβουλίου σκοπεύει να φέρουμε την Λευκορωσία εντός της οικογένειας των Ευρωπαϊκών Εθνών Σας ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλερ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Όπως είπε και ο κύριος Όστρεβίτσιους, ε, δεν είμαστε πάντα τόσο σίγουροι πως όσοι έρχονται εδώ να παρουσιάσουν κάποια πράγματα ε, δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν επιστρέφουν στη χώρα τους. Οπότε και αυτή τη φορά θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως παρακολουθούμε την κατάσταση. Γιατί είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων από το Καζακστάν που τιμωρήθηκαν αφού ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν αλλά οφείλω να σας ευχαριστήσω για την ανάλυση της ε, κατάστασης ε, και όχι μόνο ως ε, πολιτικό ακτιβιστή αλλά και ως άνθρωπο με πολιτική σκέψη γιατί λέτε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κοιτάμε και την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν πρέπει να δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αλλαγές ε, στη χώρα ή διεθνή γεγονότα όπως τους Ευρωπαϊκούς Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ιούνιο που αναφέρατε και να απαιτήσουμε συγκεκριμένες μετρήσιμες βελτιώσεις της ε, καταστάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μας είπατε πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταβάλει μια ιδιαίτερη προσπάθεια για τη Λευκορωσία και άλλες αυταρχικές χώρες για να γίνει μια κοινή πολιτική. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν δηλαδή αλλαγές, αλλά να μπορέσουμε να τις μετρήσουμε, να μετρήσουμε αυτή την πρόοδο, γιατί αυτό είναι πρόκληση. Γιατί βεβαίως ε, δεν είμαστε μόνο πολιτικό, ε, φορές ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και πολιτικός φορές και παίζουν και άλλοι παράγοντες ε, ρόλο. Τώρα να σας ρωτήσω είχατε έρθει σε μια συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν από χρόνια στην αρχή της ε, θητείας σας και συζητήσαμε και θα ήθελα να μάθω τις δυνατότητες που έχετε ε, γίνεται συζήτηση για την αλλαγή της θανατικής για την πολύ σκληρή αυτή πρακτική. Δηλαδή δεν ενημερώνουν καν τους συγγενείς πριν από την εκτέλεση να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Και βεβαίω ε, τώρα δεν υπάρχουν ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως μια συμπροεδρία γιατί η Λευκορωσία είναι πάντα στην Σύνοδο του Ιουνίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Σύνοδο του Μαρτίου. Αλλά τώρα πλέον δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες, οπότε μπορούμε να πάμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, είτε με ένα ψήφισμα ή να έρθουμε σε επαφή με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες που είναι εκεί. Και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να στηρίξουμε την παράταση της εντολής σας και θα λάβετε μια πρόσκληση για πρόσβαση στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Στρογεύσκη και μετά στους λοιπούς παρεμβαίνοντες. Η διπλωματική αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας βρίσκεται στην αίθουσα, αλλά δεν θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Της αντιπροσωπείας. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα οι καλεσμένοι μας να έχουν την ευκαιρία, ευκαιρία να μιλήσουν. Αναφερθήκατε στην μακρά εμπειρία που έχετε και αναφερθήκατε στις επιφυλάξεις σας για ορισμένες πτυχές της πολιτικής της Λευκορωσίας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά και δίνω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος και παρακαλώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Τα πολύ ουσιαστικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρέχουσα συγκυρία και η πίεση τελικά μπορεί να ασκήσει έναντι του κυρίου Λουκασέγκο. Δεδομένη τη ε, σημερινή οικονομική κρίση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου στη Λευκορωσία και δεδομένου της ε, φλέγουσας επιθυμία της ε, κυβέρνηση της Λευκορωσίας να υπάρξει παράταση των ενισχύσεων και των δανειακών συμβάσεων, των δανείων και των πιστώσεων, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία από πλευράς κυβέρνησης της ε, Λευκορωσίας να υπάρχει οικονομική στήριξη του καθεστώτος, θα πρέπει τη βοήθεια που δίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να την δίνεται εάν συνοδεύεται από δημοκρατικές αλλαγές, έτσι ώστε να υπάρξει ένα καθεστώς, ένα status quo, να μην οπισθοχωρήσουμε τουλάχιστον, να μην, να μην υποχωρήσουμε από την ε, κατάσταση και να μην γίνουμε χειρότερα αλλιώ. είδατε τι έγινε το 2008, ας σας το θυμίσω. Δάνειο τριών δις έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που βοήθησε την κυβέρνηση να, επιβιώσει, να επιβιώσει μέχρι το 2010 και τις εκλογές. Αύξησαν τους μισθούς λίγο πριν από τις εκλογές και έτσι επανεξελέγει ο πρόεδρος και τελικά ε, μετά ε, τέθηκε στο ψυγείο κάθε συζήτηση για μεταρρύθμιση. Επομένως μην πιστεύετε τα λόγια του, μην τα θεωρείτε δεδομένα τις υποσχέσεις του Πρόεδρου Λουκασέκο. Βάλτε σημεία αναφοράς, δίνετε τη βοήθεια μόνο με την εκπλήρωση ορισμένων όρων και προϋποθέσεων. Οι πολίτες της Λευκορωσίας θα πρέπει να μπορούν να μιλήσουν και να ακουστεί η φωνή τους είναι ελάχιστες προϋποθέσεις αυτές για να υπάρχει ε, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, κάτι το οποίο απουσιάζει από τη Λευκορωσία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαράστσι από τα Ηνωμένα Έθνη. Κοιτάξτε, γιατί ε, θανατική ποινή. Φέτος είχαμε μία καταδίκη και τρεις εκτελέσεις. Πέρσι ο δικηγόρος ενώ μίας από τις μητέρες που ζητούσε τουλάχιστον το σώμα, τη σωρό του εκτελεστέντος γιού για να το θάψει, την περασμένη εβδομάδα της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάδοση πορνογραφικού υλικού. Ε, ο δικηγόρος της μητέρας υπέβαλε το αίτημα η μητέρα να πάρει το ισορό του εκτελεστέντου γιού της για ε, να το θάψει. Και αυτή ήταν η απάντηση του κράτους, η εκτόξευση αυτών των κατηγοριών έναντι της μητέρας. Και αυτό μας λέει πολλά για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα αυτή. Ίσως η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει, είναι ένα one-man show, το show ε, αρχή ενός ανδρός και οι σχέσεις εξουσίας και ο αγώνας για την εξουσία ε, είναι προϊόν τόσο έντονης ε, διασύνδεσης μεταξύ της οικονομίας και των συνταγματικών διατάξεων που είναι πολύ δύσκολο να λυθεί αυτός ο γόρτιος δεσμός. Όμως διασφαλίστε ότι δεν θα επιτρέψετε στο σύστημα της Λευκορουσίας να θέσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά μέρο και να μπορέσει ε, κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών αναταράξεων πριν ή μετά να σημειώσει νίκη έναντι των εταίρων, των Ευρωπαίων εταίρων. Για παράδειγμα, ε, την εντολή των ΗΕ, την οποία εκπροσωπώ, τα δικά σας αιτήματα για τη βελτίωση της ε, κατάστασης. Μην επιτρέψετε στον πρόεδρο Λουκασέγκο να ερμηνεύσει αυτά τα αιτήματα ως διεθνείς προκλήσεις για μια καθεστική κατάσταση. Μην ε, τον ακολουθήσετε στη δική του, αν θέλετε, ατραπό για την έννοια της σταθερότητας, γιατί ε, χαρακτηρίζει σταθερότητα αυτό το οποίο είναι καταπίεση και καταστολή. Και μην το κάνετε μόνο και κλεισμένον των θυρών, αλλά και δημόσια. Μην ξεχάσετε τα ονόματα αυτών που ε, έχουν προβλήματα, ανθρώπων και οργανώσεων. Να αναφέρετε αυτά τα ονόματα ε, των ανθρώπων αλλά και των οργανώσεων. Να τα αναφέρετε δημόσια ε, γιατί έτσι στηρίζεται όλους αυτούς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αντίστασης εκ των έσω σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ θερμά. Θα παρακολουθήσουμε πραγματικά εκ του σύνεγγης την εξέλιξη της κατάστασης στη Λευκορωσία και δεδομένου ότι η διπλωματική αντιπροσωπεία της χώρας αυτής είναι παρούσα στην αίθουσα, θα θέλαμε να γνωρίζουν ότι θα ασχοληθούμε και θα ε, στενά θα παρακολουθήσουμε έτσι ώστε ο κύριος Πιαλάσκη να μην ε, υποστεί ε, καμία απειλή ή άλλου είδους δυσκολία κατά την επιστροφή του στο Μίνσκ. Θα το παρακολουθούμε στενά την άφηξή του και την παρουσία του εκεί. Ευχαριστώ.